Good afternoon, everybody. Καλησπέρα σε όλους. Να σας ε, καλωσορίσω όλους θερμά σε αυτή τη νέα αίθουσα συνεδριάσεων. Θα είναι η αίθουσα συνεδριάσεων μας για τους επόμενους τρεις μήνες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την συνεδρίασή μας, εγκρίνοντας αρχικά την ημερήσια διάταξη με μια αλλαγή κατόπιν αιτήματος ε, της εισηγήτριας κυρίας Χάρμ στο σημείο 9 το κοινοτικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια θα το εξετάσουμε αύριο, 3η 10 Φεβρουαρίου, στο τέλος του απογευματινής συνεδρίασης, γύρω στις 6 το απόγευμα. Επίσης, να σας ανακοινώσω πως έχουμε διερμηνία προς και από όλες τις γλώσσες και ότι η συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται στο ίντερνετ ε, σήμερα το απόγευμα. Το αποτέλεσμα της γραπτής διαδικασίας είναι πως οι συντονιστές συμφώνησαν για μια γραπτή διαδικασία ότι η συνεδρίαση της 16 Μαρτίου φέτος θα πρέπει να γίνει ως ήθιστε από τις 3 μέχρι τις 6.30 και ότι οι ψηφοφορίες θα γίνουν για γνωμοδοτήσεις αλλά όχι για εκθέσεις στις 5 το απόγευμα. Η συνεδρίαση της Επιτροπής λοιπόν στις 16 ε, Μαρτίου θα γίνει. Then I come to item τα πρακτικά δε των προηγούμενων συνεδριάσεων θα εγκριθούν εάν μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης δεν υπάρξουν αντιρρήσεις. Πάμε στο σημείο 4 της σημερινής διάταξης. Έχουμε τροποποίηση του κανονισμού για τη θέσπιση κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών όσον αφορά τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών. Και θα δώσω το λόγο στον ε, συντάκτη της νομοδότησης, τον κύριο Μπόκουσλαου Σόνικ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το βασικό θέμα της γνωμοδότησης είναι η αλλαγή στον ορισμό του κρέατος πουλερικών στο πλαίσιο της κοινή οργάνωσης αγοράς. Για το κρέας πουλερικών. Το κρέας πουλερικών που καταναλώνεται στα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι της καλύτερης δυνατής ποιότητας. Και αυτό προς το συμφέρον της ασφάλειας των τροφίμων θα πρέπει να διασφαλίσουμε, δηλαδή, ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν αντιμετωπίζουν κανένα κίνδυνο Ως εκ τούτου, οι αξιολογήσεις κινδύνου είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει να γίνονται προς όφελος της ε, δημόσιας υγείας. Από το 1990 έχει αυξηθεί η κατανάλωση κρέατος πουλερικών. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών. Γι' αυτό και αρχίσαμε να εξετάζουμε πιο προσεκτικά τη διαδικασία παραγωγής. Το 1997 σταμάτησαν οι εισαγωγές πουλερικών ε, από τις ίπα για λόγους ε, υγείας, λόγω της χρήσης διαφόρων χημικών στην κατεργασία του κρέατος πουλερικών. Λόγω της τεχνολογικής πρόοδου μια νέα, ένας νέος ορισμός χρειάζεται για το κρέας πουλερικών. Ε, ο ισχύων ορισμός είναι εξαιρετικά περιοριστικός και καθιστά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες αδύνατες. Το έγγραφο το οποίο εξετάζουμε ωστόσο θα μπορούσε να οδηγήσει σε νομική αβεβαιότητα, γι' αυτό και απορρίπτω το κείμενο της Κομισιόν που τροποποιεί τον κανονισμό αυτό. είναι ένα κείμενο το οποίο θέλει να καταργήσει τον ορισμό του νοπού κρέατος πουλερικών στο σημείο 5. Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε αντίφαση με το προήμιο του κειμένου. Καθώς ε, είμαι νομικός και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, στόχος της οποίας είναι να προστατεύει τη δημόσια υγεία, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να υποστηρίξουν αυτή την τροπολογία για την διαγραφή. Απ' την άλλη πλευρά, οι κτηνοτρόφοι μας χρειάζεται να πληρούν πολύ αυστηρά κριτήρια στην διαδικασία παραγωγής, καθώς και κριτήρια ευημερίας των ζώων, ενώ απ' την άλλη εισάγουμε κρέας το οποίο έχει υποστεί χημική κατεργασία από άλλες χώρες. Θα πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν τι προτιμάμε. Προτιμάμε την δική μας παραγωγή ή την χρήση χημικών. Σας ευχαριστώ κύριε Σόνικ. Έχω δύο μιλητές, τον σκιώδη συγητή από την σοσιαλιστική ομάδα, την κυρία Φερέιρα και τον σκιώδη συγγήτρια από την ομάδα Γκουε, την κυρία Λεωτάρη. Κυρία Φερέιρα πρώτα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής που διευκρινίζει ορισμένα πράγματα και επιτρέπει σήμερα να είμαστε πιο συγκεκριμένοι για ορισμένους ορισμούς. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά ποια είναι η θέση του συναδέλφου που θέλει να καταργήσει το σημείο 5, το οποίο κατά την άποψή μου επαναπροσδιορίζει τον οπό κρέας πουλερικών και θεωρώ ότι πρέπει να διατηρηθεί ο ορισμός αυτός που προτείνεται από την Κομισιόν. Εγώ θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση στην Κομισιόν σε σχέση με την πρόταση που είχε γίνει σε επίπεδο Συμβουλίου και η οποία είχε απορριφθεί το Δεκέμβριο σε σχέση με την χρήση ορισμένων ε, χλωριούχων ουσιών για την ε, Απολύμαση του κρέατος πουλερικών. Αυτή η πρόταση χρονολογείται από το Δεκέμβριο και αναφέρεται στην πρόταση κανονισμού. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν συμφωνούμε μεταξύ μας ότι η αναφορά στις πολυματικές αυτές ουσίες θεωρείται πλέον πεπαλαιωμένη και αν χρειάζεται να βρίσκεται εδώ ή όχι. Αυτή είναι η ερώτηση που έχω να θέσω προς την Κομισιόν και δεν καταλαβαίνω καλά Ποιος είναι ο στόχος ε, της τροπολογίας του συναδέλφου. Σας ευχαριστώ κυρία Φερέρα. Το λόγο έχει η κυρία Λεωτάρ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. τα πουλερικά σήμερα δεν παράγονται με γεωργικό τρόπο, κτηνοτροφικό τρόπο παραδοσιακό, αλλά με βιομηχανικό τρόπο. Δεν θα το αναλύσω αυτό περισσότερο, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό το ότι γίνεται διαφήμιση και χορηγεί, λαμβάνει χορήγηση και ε, επιδότηση στην Ολλανδική τηλεόραση για να προωθηθεί η κατανάλωση του κρέατος πουλερικών. Όταν βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση της βιομηχανίας και βλέπουμε ε, το γεγονός ότι χρειάζεται να χρησιμοποιούμε, να, καταναλώνουμε αυτά τα πουλερικά, τα οποία υπόκειται σε μια διαδικασία απολύμασης στη ΣΥΠΑ, γιατί δεν έχουμε αρκετό κρέας πουλερικών εδώ. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ε, γίνεται κάτι τέτοιο. Τώρα, αν ε, η τροπολογία του εισηγητή σημαίνει πως οι καταναλωτές θα αγοράζουν νοπό κρέα πουλερικών το οποίο έχει υποστεί αυτή τη διαδικασία απολύμασης αν ο στόχο είναι να αποφύγουμε κάτι τέτοιο το υποστηρίζω γιατί νομίζω το νοπό σημαίνει κάτι συγκεκριμένο και πρέπει ο ορισμό να είναι ξεκάθαρο. σω λοιπόν ο εισηγητή να πρέπει να μα πει κάτι γι' αυτό αν ο στόχο είναι αυτό λοιπόν τον υποστηρίζω Σα ευχαριστούμε κυρία Λεωτάρ ο κύριος Χόπενστέτ Ja, vielleicht nur ein ganz kurzer Beitrag. Ich habe Πολύ σύντομα. Δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με την πρόταση αυτή, διότι είχα άλλες δουλειές και δεν είχαμε πολύ χρόνο, αλλά ως προς τη βασική αρχή θα πρέπει να προσέξουμε το γεγονός ότι έχουμε στην Ευρώπη και στις διάφορες χώρες ε, κανόνες ε, υγιεινής. Ε, για όλες ε, τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τα πουλερικά. Υπάρχουν ε, εξειδικευμένες διαδικασίες, όχι μόνο βιομηχανικές, αλλά και γεωργικές. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, δεν παίζουν ασήμαντο ρόλο στις ε, εγχώριες αγορές. Ε, θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε να μην εξισώσουμε όλα. Θα πρέπει να προσέξουμε τις μεθόδους σφαγής. 25 χρόνια εργάστηκα στον τομέα των πουλερικών. Γνωρίζω πολύ καλά πώς λειτουργούν τα πράγματα σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Ε, ξέρουμε τους αυστηρούς ε, κανόνες υγιεινής ε, που εφαρμόζονται ξέρουμε τις μεθόδους αναισθητοποίησης πριν τη σφαγή. Στην Ευρώπη έχουμε πολύ ψηλά πρότυπα, στη Γαλλία, στη Γερμανία. λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο πραγματοποιούνται τα πράγματα παντού. σημαντικό είναι να Ε, τηρούνται οι κανόνες ε, και από όλους ε, τους προμηθευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για σαφείς κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται και προς συμφέρον του καταναλωτή αλλά και για την προστασία των ζώων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χόπενστεντ. Ο κύριος Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο για την γνωμοδότησή του. Θα ήθελα να θέξω μόνο ένα θέμα. Γιατί όταν διαβάζουμε αυτή τη φράση έγκριση χρήση ορισμένων ουσιών για την απολύμανση των κρέατος πουλερικών, με κάνει να θυμηθώ το μάχη που δώσαμε πριν από κάποιους μήνες για την εισαγωγή, το, τις εισαγωγές ε, κρέατος πουλερικών από την Αμερική. Και αυτό γιατί από ό,τι θυμάμαι βουτάνε τα, βαφτίζουν τα κοτόπουλα <laughs> στη χλωρίνη. Και μετά το βουτάνε και στις ε, σάλτσες του Kentucky Fried Chicken. Ε, ακόμα και το ίδιο το κεντάκι fried chicken θα ήταν λόγος για να απαγορέψουμε τις αγωγές ε, πουλερικών από τις ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, ε, εγώ θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε, να μου επιβεβαιώσει μάλλον ο φίλος εδώ αλλά και η Κομισιόν ότι τίποτα σε όλα αυτά δεν θα ανοίξει την πόρτα στα χλωριωμένα κοτόπουλα, είτε σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση από τους Αμερικανούς. Μην τυχόν μας πούνε δηλαδή ότι εμείς βάζουμε άλλες ουσίες, γιατί να μην βάλουν και αυτοί λίγο χλώριο. Αυτά λοιπόν, αν μου το αποψαφνίσετε αυτό δεν έχω πρόβλημα. <clears throat> Ευχαριστώ τον Τζον ε, Πόουις Ολοκληρώσαμε τον ε, κατάλογο των ομιλητών. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Στο πρόγραμμά μου λέει ότι εκπρόσωπος της Κομισιόν, κύριος Λούντα, έχετε το λόγο. Okay, excusez Um... Ναι. Όσον αφορά το θέμα της ε, κατεργασίας με χλώριο και για να απαντήσω στις ερωτήσεις που ετέθησαν, η Κομισιόν σαφώς ε, ε, υποδεικνύει ότι στην περίπτωση που η πρόταση της Κομισιόν που, επιτρέ που επιτρέπει τη χρήση αυτών των νησιών δεν εγκριθεί, θα αποσύρουμε τον ορισμό από την πρόταση αυτή και περί αυτού πρόκειται. Και υπάρχει θέμα διαδικασίας θα έλεγα, διότι για να κερδίσουμε χρόνο υποβάλαμε την πρόταση όσοι έχει στο Συμβούλιο και στο Συμβούλιο θα πρέπει να αποσύρουμε το κομμάτι που αφορά την αλλαγή του ορισμού του νοπού κρέατος ώστε να επιτρέπεται η κατεργασία με αυτές τις ε, ουσίες. Ε, θα το αποσύρουμε λοιπόν αυτό, άρα λοιπόν οι ουσίες αυτές δεν θα επιτρέπονται. Ελπίζω να ήμουν σαφής. Έπειτα, υπήρχε το θέμα το αν θα αποσύρουμε ή όχι το σημείο 5. 2-5 που αφορά την αποσαφήνιση του ορισμού των ε, παρασκευασμάτων με βάση νοπό κρέας πουλερικών. Η Κομισιόν δεν κατανοεί για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η πρόταση. Άκουσα τον κύριο Σόνικ που σωστά μα είπε για την καλύτερη δυνατή ποιότητα και ακριβώ κύριε Σόνικ η πρότασή μα προ αυτήν την κατεύθυνση ε, πηγαίνει γιατί θα αποφύγουμε τον παραπλανηθούν οι καταναλωτές. Γιατί λέμε ότι κάθε ε, παρασκεύασμα με βάση νοπό κρέας πουλερικών απαραίτητο θα πρέπει να περιέχει νοπό κρέας. Και δεν είναι δυνατόν να αποψύχεται και έπειτα αυτό το κρέας να πωλείται ως νοπό κρέας και να παραπλανεί τον καταναλωτή. Ακριβώς λοιπόν προς χάρη ε, ποιότητας είναι απαραίτητο να εισαχθεί αυτή η αποσαφήνιση όσον αφορά τα παρασκευάσματα με βάση νοπό κρέας πουλερικών. Και έπειτα ετέθηκε η ερώτηση του αν οι θα μπορούσαν να μας πάνε σε πάνελ. Νομίζω πως την ερώτηση θα πρέπει να την υποβάλουμε στους Αμερικανούς. Εγώ θα μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις οι Αμερικανοί για να δουν ακριβώς εάν είναι σκόπιμο να ξεκινήσουν και πάλι ένα νέο πάνελ. Ελπίζω να απάντησα έτσι στις διάφορες ερωτήσεις. Διαφορετικά ε, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τώρα δώσουμε το λόγο στον κύριο Σόνικ. E, Κύριε Πρόεδρε, είδα ότι ο πρόσωπο τη Επιτροπή αναφέρθηκε σε αυτή την ε, κατάσταση, γιατί μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο μεταβάλλεται αυτή τη στιγμή, οπότε τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Και μάλιστα είχαμε και αυτή την αλλαγή στην οποία αναφέρθηκα που ε, ήρθε στις 19 Δεκεμβρίου. Κοιτάξτε, εγώ τοποθετήθηκα. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον ορισμό του νοπού κρέατος και να ε, βάλουμε αυτή τη δυνατότητα χρησιμοποίησης χημικών ουσιών. Αυτό θέλω να πω. Εάν η Επιτροπή μπορεί να μου εγγυηθεί ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία, χωρί πρόβλημα. Αυτή πάντω είναι η πρόθεσή μα. Αν η Επιτροπή μα διαβεβαιώνει ε, για το ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, τότε εντάξει. Και ο ίδιο ε, ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή είπε ότι υπάρχει πρόθεση τροποποίηση του κανονισμού ε, για να, στο μέλλον για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σόνικ. Και τώρα ολοκληρώσαμε τη συζήτηση στο θέμα αυτό. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι σήμερα. 9 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα. Και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 17 Φεβρουαρίου. Και μετά θα υποβληθεί στην Επιτροπή Γεωργίας η ψηφοφορία στην 31η Μαρτίου και θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Απριλίου. Ωραία. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη συζήτηση για το θέμα αυτό και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη έκθεση ε, στην κυρία Μούρκο και θα της δώσουμε το λόγο για να παρουσιάσει το θέμα της προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Κυρία Μούρκο, έχετε το λόγο. Mr. Chair. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συγγνώμη, διακόπτη Πρόεδρος. Ο κύριος Μπόης ε, ε, θέλει να τοποθετηθεί από τι διαδικασίε. Μάλιστα, συγγνώμη, λέει κυρία Μούρκο, δεν τον είδα. Ζητώ συγγνώμη από την εισηγήτρια. Απλά και μόνο θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να πω για το θέμα αυτό, ότι πιστεύω ότι να μιλάτε για προθεσμία για υποβολή τροπολογιών πριν καν από τη λήξη τη σημερινή συνεδρίαση ε, είναι κάτι παράλογο. σω θα μπορούσε να δοθεί μια παράταση για μία-δύο ημέρε. και θα είμαστε, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ε, θα έχουμε έτοιμη την ε, γνωμοδότησή μας. Αλλά κοιτάξτε, νομίζω ότι το γεγονός ότι συζητήσαμε τώρα και βεβαίως Ε, ε η κυρία Μούρκο θα μα παρουσιάσει το επόμενο θέμα. Ε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον, θα την παρακολουθήσουμε. Τώρα να μα δείτε παράλληλα, να σκεφτόμαστε και τι απόψει μα και μέχρι τι 6 να σα έχουμε υποβάλει. Τι να σα πω, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι κάπω υπερβολικό. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να ψηφίσουμε στις 17 Φεβρουαρίου. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να πάμε στις 16 Μαρτίου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Η Επιτροπή Γεωργίας πότε θα ψηφίσει? Κυρία Μούρκο, ήθελα να πω δύο λόγια ε, ε, για να εξηγήσω και το γιατί δουλεύουμε κάτω από τόσο ασυνήθιστες συνθήκες και γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα. Και έχουμε και την προθεσμία και τις ερπολογίες σήμερα πάλι. Η προθεσμία για την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας, που είναι η αρμόδια επιτροπή επί της ουσίας, είναι η 18η Μαρτίου. Αν λοιπόν δεν. Ε, ε, αν ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα και όχι. Όχι, σα συγγνώμη. Φεβρουάριο, Φεβρουάριο διορθώνει η μιλήτρια. Δεν πρόκειται να λάβει υπόψη τη ε, η Επιτροπή Γεωργία απόψη μα. Κύριε Πόση, συγγνώμη. Μα μόλι είδα το φάκελο και φαίνεται ότι θα ψηφίσει τι 30-31 Μαρτίου η Επιτροπή Γεωργία. Uh, ε, for... Προθεσμία για, για τις εκθέσει των εισηγητών να το πω διαφορετικά. Τα πράγματα έχουν ω εξή. Για να, ληφθεί υπόψη, να ληφθούν υπόψη οι απόψει μα, πρέπει να έχουμε συζητήσει και να έχουμε μέχρι τότε. Καταλαβαίνω ότι η Επιτροπή περιβάλλοντο. Ε, μάλλον καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο παρά να ψηφίσουμε σήμερα. Τώρα πρέπει να σα πω στην Επιτροπή Περιβάλλοντο. Πρέπει να σα πω ότι και εγώ αισθάνθηκα ιδιαίτερα άβολα αναγκάστηκα να συντάξω το σχέδιο γνωμοδότηση μέσα σε δύο ημέρε την περασμένη εβδομάδα. Και πράγματι είναι ασυνήθιστε αυτέ ε, οι συνθήκε εργασία. Βεβαίω ε, ε, αναγκάστηκα να συμμορφωθώ κάτω από αυτέ τι δύσκολε περιστάσει. Λοιπόν, να προτείνω το εξή. Δεν θέλω να καθυστερήσω τη τώρα. Αφήστε όμω τη δική μου ιδέα. Να δούμε, να δούμε. Μήπω μπορούμε να βρούμε λίγο περισσότερο χρόνο. Πέραν τη έκτη απογευματινή σήμερα. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Εάν η βασική επιτροπή δεν ψηφίζει πριν την 31 η Μαρτίου και έχουμε και την εδώ ψηφίσει 16, γιατί δεν το κάνουμε αυτό, μα έχουμε το χρόνο. Τώρα θα έχουμε όλο τον χρόνο να βάλουμε τι προτάσει μα. Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω. When we have all the amendments in English. Έχουμε όλες τις απολογίες στα αγγλικά, άρα αύριο. Δεν γίνεται αύριο. Αύριο το μέχρι το μεσημέρι στις 12. Κύριε Τζάξον. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να μιλήσω. Πού, πού μιλάω μάλλον. Α, εδώ, ωραία. Θα βοηθούσε αν είχαμε προθεσμία μέχρι αύριο. Αλλά να πω το εξή. Θα έπρεπε η Επιτροπή μα να έχει εκφράσει αντιρρήσει τη και ίσω και ακόμα και τώρα υπάρχει χρόνο να εκφράσουμε ε, τι αντιρρήσει μα, γιατί δεν είμαστε η αρμόδια επιτροπή. Καταλαβαίνω ότι το θέμα τη κατάσταση των ζώων και τη ευζοία είναι αρμοδιότητα τη Επιτροπή Γεωργία, αλλά στην ουσία εμεί είμαστε υπεύθυνοι, νομίζω, για τι ε, δοκιμέ στα καλλιντικά. Και αν δείτε το άρθρο 2 τη οδηγία ε, με εισηγήτρια την κυρία Μόρκο αναφέρεται ότι η οδηγία δεν θα ισχύσει σε γεωργικές πρακτικές, πρακτικές ε, που γίνονται για την ε, ε, αναγνώριση της εκτροφής των ζώων, αναγνώριση των ζώων κτλ. Άρα λοιπόν δεν αναφέρεται στα θέματα για τα οποία είναι αρμόδια η Επιτροπή Γεωργίας. Και εμεί είμαστε η αρμόδια επιτροπή για περιβάλλον, δημόσια υγεία και ασφάλεια τροφίμων. Μα γιατί λοιπόν δίνουμε ε, την οδηγία αυτή στην Επιτροπή Γεωργία. Εμεί είμαστε υπεύθυνοι και νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία. Να εκφράσουμε τι αντιρρήσει μα, αποστέλετε μια επιστολή στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και πραγματικά, πραγματικά να εκφράσουμε αντιρρήσεις. Γιατί μα αναγκάζουν βεβαιασμένα να εκφράσουμε τι απόψει ενώ θα έπρεπε να... Α, με βλέπω και στην τηλεόραση, λέει η κυρία Τζάξο, δεν το καταλάβει ότι με δείχνει. Ε, άρα λοιπόν, τουλάχιστον ε, θα έπρεπε να ζητήσουμε διεύρυνση προθεσμίας. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από εσά, κύριε Πρόεδρε, κατά πόσο μπορείτε να έρθετε σε επαφή με του συντονιστέ ε, ε, και τους ε, υπεύθυνου των άλλων ομάδων για να αποστείλουμε μια επιστολή στο πρόεδρο του Κοινοβουλίου να πούμε ότι έγινε λάθος όσον αφορά την, τον καθορισμό τη αρμόδια επιτροπής και να ζητήσουμε να φύγει τελείω από την ημερήσια διάταξη αυτού του Κοινοβουλίου. Με την καινούργια θητεία, νομίζω το Κοινοβουλίο θα δει τα πράγματα με ένα άλλο μάτι και θα στείλει το θέμα αυτό στην αρμόδια επιτροπή. Τι λέτε για αυτή μου την ιδέα. Jackson. Maar gelijk krijgen κύριε Τσάξον, ε, έχετε δίκιο, πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, ζήτησε ενισχυμένη συνεργασία, αλλά απορρίφθηκε αυτό. Θα μπορούσαμε να ανακοινήσουμε πάλι τη διαδικασία, αλλά μάλλον δεν θα πετύχουμε τίποτα. Νομίζω ότι έχετε δίκιο ότι λάθος δόθηκε αυτή στην Επιτροπή Γεωργία και είναι λάθος που δεν έχουμε διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα τώρα. Ελπίζω το επόμενο κοινοβούλιο να μπορεί να χειριστεί με καλύτερο τρόπο τα θέματα αυτά, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι μια αναβολή τώρα θα ήταν σωστή, διότι έχει ληφθεί απόφαση και πρέπει να τη δεχτούμε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ε, σε προθεσμία αύριο το μεσημέρι. Δίνω το λόγο στην κυρία Μούρκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λογική είναι η πρότασή σας, αν και συμφωνώ ότι θα έπρεπε να, δοθεί, θα έπρεπε να έχει δοθεί έκθεση αυτή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η διάσκεψη των Προέδρων όμως έλαβε απόφαση. Μου ζητάτε να παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης. Και μπορώ να πω ότι είναι καιρός για αναθεώρηση της παλιάς οδηγίας του 1986. Η κυρία Κάρολαϊν Τζάκσον ήταν η συγγήτρια τότε. Από ό,τι γνωρίζω όμως ήταν μια από αυτούς που 10 χρόνια αργότερα ε, απέτησαν αναθεώρηση της οδηγίας αυτής. Η πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει την εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Ευρώπη και την προσέγγιση της ε, ε, της έννοιας της προστασίας των ζώων ε, στα επιστημονικά πειράματα. Σκοπός είναι να προταθούν εναλλακτικές λύσεις ε, στις δοκιμές σε ζώα και έχουμε τις ε, τρεις βασικές αρχές, την αντικατάσταση, την εξέλιξη και τη μείωση της χρήσης των ζώων. Υποχρεωτική χρήση μεθόδων που να ακολουθούν τις τρεις αυτές αρχές αποτελούν βήμα προόδου σε σχέση με την ε, λιγότερο αυστηρή νομοθεσία στην οδηγία του 1986. Ζωτικής σημασίας ε, είναι και ε, ο καθορισμός του ανώτατου ορίου του πόνου για τα ζώα κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Δεν θα πρέπει να, να επιτρέπονται δοκιμές ε, που προκαλούν ε, ε, έντονο πόνο στα ζώα. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι στόχοι με την πρόταση αυτή. Ως συντάκτρια της γνωμοδότησης, επικροτώ την πρόταση της Κομισιόν. Περιέχει μέτρα που βελτιώνουν την προστασία των ζώων και εισάγει αυστηρούς κανόνες που ακολουθούν διεθνώς αποδεκτές αρχές σωστών επιστημών πρακτικών. Αναφέρονται ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των ζώων ε, για επιστημονικούς σκοπούς. επικροτώ τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας που περιλαμβάνει ε, ασπόνδυλα ζώα καθώς ε, και ε, ε, έμβρια ζώων που αισθάνονται. Επίσης την εισαγωγή μη βάναυσων τρόπων θανάτωσης στις διαδικασίες αυτές. Ένα από τα βασικά σημεία είναι η χρήση μη ανθρώπινων πρωτευόντων θηλαστικών που θα πρέπει να μειωθεί βαθμιαία με άμεση απαγόρευση των μεγάλων πυθικοειδών. Η βαθμιαία μείωση των ε, πρωτευόντων θηλαστικών αυτών Δηλαδή τα παιδιά ε, πρωτευόντων θηλαστικών ε, που έχουν ε, ε, συλληφθεί στην ε, φύση και είναι σημαντική αυτή η απαγόρευση ε, και για ηθικούς λόγους. Το μέτρο αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα ε, μειώσει την πίεση στα, στους άγριους πληθυσμούς και θα αποτρέψει την, τη βάναυση μεταχείριση των ζώων αυτών. Σε αντίθεση όμως με την πρόταση της Κομισιόν πιστεύουμε ότι εξαιρέσεις στον ότι μια εξαίρεση που βρίσκεται στο άρθρο 35 θα αφήσει ανοιχτό ένα παράθυρο για ε, δοκιμές σε εργαστήρια αυτών ε, των ε, απειλούμενων ειδών. Η ρήτρα εξασφάλισης για τα μεγάλα πυθικοειδή κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να διαγραφεί. Η αυτό συνάδει με τις ε, ανησυχίες που ε, εκφράζονται στην οδηγία του 86, πάνω από 20 χρόνια πριν η, χρήση των, ε, των, ε, η υπαγόρευση της χρήσης των ε, μεγάλων πυθικοειδών ήδη εφαρμόζεται σε κάποια κράτη-μέλη. Η γρήγορη αναρμόνιση σε όλη την Ευρώπη είναι κατά τη γνώμη μας δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Στην πρόταση θα θέλαμε να δούμε κατηγοριοποίηση των διαδικασιών Υπάρχει έλλειψη κριτηρίων για την κατηγοριοποίηση των διαδικασιών και προτείνουμε ένα νέο παράρτημα ε, για την ε, κατηγοριοποίηση της, ε, για τον καθορισμό της ε, σοβαρότητας των διαφόρων διαδικασιών. Συζητήσαμε το θέμα και ανακαλύψαμε ότι διάφορες δράσεις ήδη έχουν ξεκινήσει. Ο καθορισμός ε, λοιπόν ε, της ε, σοβαρότητας σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή που υπάρχει στην πρότασή μας θα είναι μεταβατικό μέτρο και θα προκαλέσει σύγχυση στα κράτη-μέλη όπου ήδη εφαρμόζεται μια τέτοια κατηγοριοποίηση. Σας καλώ λοιπόν να επιδείξετε κατανόηση. Θα αποσύρουμε το σχετικό παράρτημα. διότι όπως είπα, θα υπάρξει επικάλυψη των προσπαθειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο προς το παρόν. Μου είπαν όμως ότι σε 18 μήνες θα είναι έτοιμη η κατηγοριοποίηση ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να τονίσω και τις ε, αρχές στο κεφάλαιο 4 της πρότασης που έχουν να κάνουν με τη δεοντολογία. Πιστεύουμε ότι είναι βασικό χαρακτηριστικό της πρότασης. Ξέρουμε ότι Αναθεώρηση γίνεται τακτικά σε 21 κράτη-μέλη. Θα πρέπει όμως ε, να αποτελέσουν βασικό μέρος ε, της ε, διαδικασίας πιστοποίησης. Θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση της βλάβης και του ωφέλους που ζυγίζει την ε, χρήση των ζώων σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επίσης, ε, μια τέτοια αξιολόγηση θα ενθαρρύνει την ε, σωστή επιστήμη, καθώς, όπως άλλωστε και οι τρεις αρχές που αναφέραμε, της μείωσης, της αντικατάστασης κλπ. Οι κυρίες που κάθονται δίπλα μου που είναι συνεργάτες μου ε, ε, επικροτούν τις ε, εθνικές επιθεωρήσεις. Κατ' ελάχιστον μία το χρόνο. Πιστεύουμε ότι η ιδέα αυτή θα μπορούσε να ενισχυθεί. Θα θέλαμε λοιπόν και υπέβαλα σχετική τροπολογία να υπάρξει η δυνατότητα ευρωπαϊκής επιθεώρησης ώστε επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να κάνουν επιθεωρήσεις χωρίς προειδοποίηση, ώστε να ε, διασφαλίζουν την ε, σωστή και ενιαία εφαρμογή των κανόνων στα κράτη-μέλη. Κατά τη γνώμη μου, η διαφάνεια αποτελεί μια από τις αρχές που θα πρέπει να ενισχυθούν. Γνωρίζουμε ότι πραγματοποιείται πολύ ε, βασική έρευνα στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά πειράματα δεν είναι τόσο διαφανή όσο άλλα. Τώρα λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε υποχρεωτικούς τους σχετικούς κανόνες. Επίσης, όσον αφορά τις εκθέσεις και τα αποτελέσματα των ερευνών, θα πρέπει να δημοσιεύονται. Γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημασία των εμπιστευτικών πληροφοριών. Υπάρχουν μέρη της πρότασης που καλύπτουν ε, το συγκεκριμένο θέμα. Εμένουμε στην αρχή αυτή. Θα θέλαμε όμως να είναι απαραίτητα λιγότερα πειράματα σε ζώα. Τη στιγμή που ήδη υπάρχουν σχετικά αποτελέσματα ερευνών σε άλλους τομείς. Η ανταλλαγή στοιχείων και η χρήση στοιχείων που έχουν προκύψει από άλλα πειράματα θα πρέπει να μειώσουν την ανάγκη για πειράματα σε ζώα. μπορεί η Περιβαλλοντική Επιτροπή να συνεισφέρει στην πρόταση της Κομισιόν. Προτείνουμε διάφορες τροπολογίες που τονίζουν και ενισχύουν το, το βασικό πεδίο εφαρμογή ε, της πρότασης. Θα πρέπει να παρέχουμε τις ε, συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί η επιστήμη να ανθίσει, να αναπτυχθεί και θα πρέπει η αντικατάσταση των πειραμάτων ε, με ζώα να ε, βρίσκονται ε, στη βάση της πρότασης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μούρκο. Στον κατάλογό μου έχω 7 ομιλητές. Ο κύριος Χόπενστέτ, η κυρία Λιωτάρ, Τζάκσον, Γκροστέτ, και Ούμερ. Δίνω λοιπόν το λόγο στον σκιώδο εισηγητή του ΕΛΚ, τον κύριο Χόπενστέτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να καταστήσω σαφές, ε, αυτό υπόθηκε για τον κύριο Πόβης και άλλους, η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να έχει μοιραίες συνέπειες ε, για το αποτέλεσμα. Ε, σήμερα στις 11 λάβαμε το, την πρόταση της κυρίας Μούρκο. Αναβλήθηκε η προθεσμία από σήμερα στις 6 μέχρι αύριο. Αυτό σίγουρα μας βοηθάει. Αλλά δεν ε, βρισκόμαστε απλά σε μια κλειστή αίθουσα και εργαζόμαστε μεταξύ μας. Ε, βρισκόμαστε και στο μάτι της δημοσιότητας. Ε, της, ε, του τομέα των ερευνών ε, και άλλων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα που συζητάμε. Η πρόταση βασίζεται στην οδηγία του 86 θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε την πρόταση αυτή στα τέλη του 2009, το 2010, αλλά τέλος πάντων. Επικροτώ την αναθεώρηση της οδηγίας και... Έχω τις ε, τροπολογίες μου ε, στα γερμανικά, 33 τροπολογίες είναι, το Σαββατοκύριακο τις μεταφράσαμε κιόλας ε, και ε, έχουν να κάνουν ε, με αυτά που, ε, που προτάθηκαν από την Κομισιόν. Δεν ε, θα ασχοληθώ με τις επιμέρους διαδικασίες, θα το κάνουμε αυτό όταν έχουν υποβληθεί όλες οι τροπολογίες. Επί της αρχής λοιπόν επικροτούμε την τροποποίηση της παλιάς οδηγίας. Από το 1986 έχει αναπτυχθεί πολύ ο τομέας ε, των ε, πειραμάτων σε ζώα. Ως εκτινίατρος έχω ε, συλλέξει πολύ πείρα στο θέμα αυτό. Έχει καθυστερήσει πολύ η τροποποίηση της οδηγίας πρόταση αυτή στηρίζεται στις νέες γνώσεις για την προστασία των ζώων, ε, τονίζει την κατάρτιση των ε, εργαζομένων και αναφέρεται και στις ε, αρχές αυτές το τριπλό R, δηλαδή την αντικατάσταση, την μείωση και την εξέλιξη των μεθόδων. Και είτε τα πειράματα αυτά γίνονται στα πανεπιστήμια ή σε φαρμακευτικές εταιρείες. Αν δει κανείς σε ποιοι επαγγελματίες ε, εργάζονται εκεί και υπό ποιες ε, συνθήκες, σίγουρα θα έχει πολύ σεβασμό για τη δουλειά αυτή. Το υψηλό επίπεδο προστασίας ε, των ζώων θα πρέπει να ζυγιστεί σε σχέση με ε, το όφελος για τη δημόσια υγεία και η ανάπτυξη των ε, νέων φαρμακευτικών προϊόντων δεν θα πρέπει να διακυβευτεί. Ε, ως ασθενείς οι ασθενείς, όποιος θέλει να θεραπευτεί, περιμένει ε, ακριβώς ε, αυτό. Από την πρόταση της Κομισιόν ε, κατέστη σαφές ότι θα πρέπει όλα αυτά να βασίζονται σε σαφείς επιστημονικές αρχές και δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν ε, περιτά εμπόδια για ε, την έρευνα. Ε, στηρίζω τις, τα μέτρα αυτά, την εξέβρεση εναλλακτικών μεθόδων όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικέ μέθοδοι σήμερα τουλάχιστον, δεν ξέρουμε μεθαύριο τι θα γίνει. Ε, στηρίζω οτιδήποτε ε, βελτιώνει τις ε, συνθήκες των, στα πειράματα. Επίσης, η πολλή γραφειοκρατία που θα πρέπει Επίσης η πολλή γραφειοκρατία θα πρέπει να εξαλειφθεί χωρίς αυτό να επιδεινώσει την προστασία των ζώων. Η αναθεώρηση θα πρέπει να προβλέπει μία ε, διαδικασία ε, χωρίς ε, γραφειοκρατικό άχθος. Η αναθεώρηση επίσης θα πρέπει να ε, επιδιώξει εξομοίωση των κανόνων εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Δεν είναι μόνο το θέμα της προστασίας των ζώων, αλλά πρόκειται και για έναν σημαντικό τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Μια σημαντική δραστηριότητα για την ευρωπαϊκή οικονομία την έρευνα δηλαδή. Πιστεύω ότι η πρόταση αυτή θα συμβάλλει ώστε σε επίπεδο κρατών μελών να βρεθούν ε, κανόνες και μέτρα που να μπορούν να ισχύουν ε, για τα ε, πειράματα σε ζώα σε όλα τα κράτη-μέλη. Θέλουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να ανταποκρίνεται στις συνθήκες. Δεν ε, θέλω να αναφερθώ στο θέμα των πρωτευόντων θηλαστικών. Αυτό ρυθμίζεται εδώ πέρα. Ε, πρόκειται πιθανότατα για αυστηρή ε, μεταρρύθμιση αλλά ε, αναφέρθηκε το κυνήγι των ε, ζώων αυτών ε, στη φύση, το οποίο ήδη έχει απαγορευτεί. Αναφερόμαστε στην γενιά F1 και F2, τα παιδιά δηλαδή των ζώων αυτών που έχουν συλληφθεί στην Δύση. Εγώ προέρχομαι από το Ανόβερο, ε, ε, δεν ε, θα πρέπει να διακυρωθεί η κατάσταση ούτε στο Ανόβερο από το οποίο προέρχομαι, ούτε στην Ευρώπη όμως θέλουμε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των κέντρων ερευνών θα πρέπει να φροντίσουμε να μην ε, σαμποτάρουμε προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Όλα τα κέντρα ερευνών, τα πανεπιστήμια, οι επιχειρήσεις ε, βιοτεχνολογίας ε, κλπ. Ε, θα πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν νέε φαρμακευτικές ουσίε. Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στου στόχου τη οδηγία, ε, την ανταγωνιστικότητα τη ε, Ευρώπη και τι καινοτόμε θεραπευτικέ μεθόδου. Είναι σημαντικό και σε παγκόσμιο επίπεδο να προβάλλουμε πρότυπα τα οποία να ακολουθήσουν και άλλοι. Εάν ε, ασχοληθούμε μόνο με τα πρότυπα εντός της Ευρώπης, τότε πολύ σύντομα θα δούμε μεταφορά των πειραμάτων εκτός Ευρώπης και δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ήδη υπόθηκε ότι θέλουμε αξιόπιστες εναλλακτικές μεθόδους. Ε, αυτό αποτελεί μια απέτηση προς την επιστήμη, αλλά και την επιστήμη θα την ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Όποιος ε, έχει ε, δει τα πειράματα που γίνονται στα εργαστήρια, ε, θα γνωρίζει πόσο υψηλά είναι τα πρότυπα, διότι άλλωστε είναι πολύ ακριβές οι δοκιμές αυτές και οποιοδήποτε θα αναζητούσε και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Ε, κάτι που παλιά γινόταν σε ζώα τώρα γίνεται με καλλιέργεια ε, σε κύτταρα από ε, έμβρια χάμστερ αυτό και στοιχίζει λιγότερο και πρόκειται για καλό παράδειγμα πώς μπορεί να τροποποιηθεί η μέθοδος πειραμάτων σε ζώα προς το καλύτερο. Σας παρακαλώ να εξετάσετε τις τροπολογίες μου. Ε, πιστεύω ότι λαμβάνουν υπόψη την προστασία των ζώων αλλά και τις ανάγκες ε, του σχετικού τομέα. Και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε μια ε, εντελεχή συζήτηση σχετικά με τις επιμέρους προτάσεις. Ε, αυτά είχα να πω σχετικά με το τι προσπαθώ να, να πετύχω με τις τροπολογίες μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ δώσουμε το λόγο τώρα στην κυρία Φεραίρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ πιο σύντομη. Πιστεύω ότι όλοι εδώ συμφωνούμε στο ότι ε, απαιτείται η αναθεώρηση της οδηγίας που, έχει, που ε, ξεκίνησε πριν από πάνω από δύο δεκαετίες. Όλοι συμφωνούμε στο ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό και τα πειράματα με ζώα σε όλες τις χώρες και σε όλους τους πολίτες ε, δημιουργούν έντονα συναισθήματα. Νομίζω ότι και εδώ στην Επιτροπή μας όλοι επιδεικνύουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στο ε, θέμα αυτό που έχει να κάνει με το μέλλον των ζώων και με τη χρησιμοποίηση των ζώων, κυρίως των πρώτων ε, στο θέμα αυτό των πειραμάτων. Πέραν όμως των συναισθημάτων θα πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ε, ότι ε, οι Ευρωπαίοι ερευνητές ε, μπορούν να ε, προσφεύγουν στα πειράματα με τα ζώα ε, για σαντιστικούς σκοπούς, κυρίως όταν πρόκειται για πρωτεύοντα. Και γνωρίζουμε εξάλλου ότι ένας ορισμένος αριθμός πειραμάτων είναι απαραίτητος και θα πρέπει να γίνεται στα πρωτεύοντα όσον αφορά τα φάρμακα για παράδειγμα. Φάρμακα για ασθένειες όπως το AIDS, όπως η νόσος του Alzheimer, ε, η, το Parkinson, ορισμένα εμβόλια κτλ τα πειράματα αυτά είναι απαραίτητα και πρέπει να γίνουν σε πρωτεύοντα. Νομίζω επίσης ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε και το εξής. Εφόσον υποβάλλουμε προτάσεις ε, πολύ περιοριστικές, θα πρέπει να αναρωτηθούμε και το εξής για τις επιστημονικές συνέπειες ε, των προτάσεών μας και για, ε, την ε, επιστημονική τεκμηρίωση των διατάξεων που εμείς επιθυμούμε να υιοθετήσουμε. Προσωπικά πρέπει να σας πω ότι δεν έχω ε, απαραίτητα στοιχεία για το θέμα αυτό, αλλά πρέπει να σας πω ότι ε, με πλησίασαν πολλοί εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων που έχουν ορισμένες ανησυχίες ε, για το μέλλον της ε, επιστημονικής έρευνας. Και όπως είπε και ο προλαλής σας, βεβαίως ε, πρέπει να ενισχυθεί το πλαίσιο αναφοράς και ο κανονισμός, ε, η νομοθεσία γενικότερα για τα πειράματα και βεβαίως ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, ότι τα πειράματα αυτά γίνονται σε άλλες χώρες και εκεί η ρύθμιση είναι πολύ λιγότερο αυστηρή από ότι έναντι τη ρύθμιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αισθάνομαι ανησυχία, αυτό θέλω να πω. Κανείς βεβαίως δεν θέλει να βασανίζονται τα ζώα, Κανείς δεν θέλει τα ζώα να, να ε, υφίστανται αυτές τις συνέπειες στα εργαστήρια. Αλλά πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, μήπως τελικά η επιστήμη χρειάζεται αυτά τα πειράματα. Εντάξει, να ενισχύσουμε την νομοθεσία, αλλά να είμαστε και μέσα στα πλαίσια του λογικού και του εφικτού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Φερέρα, κυρία Λεωτάρ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. και ευχαριστώ την κυρία Μούρκο για την εισήγησή της. Συμφωνώ μαζί σας ότι εσείς θα έπρεπε να είστε αρμόδια από της ουσίας, αλλά μας περιπτώσει αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σε τρία σημεία σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξουν δεσμευτικοί στόχοι για τον περιορισμό των πειραμάτων σε ζώα και εκεί όπου υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις να είναι υποχρεωτικές να είναι υποχρεωτική η χρήση τους και πιστεύω πως θα πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για να αναβρεθούν εναλλακτικέ λύσεις διότι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 12 εκατομμύρια πειραματόζωα χρησιμοποιούνται ή μάλλον γίνεται κατάχρηση αυτών. Συζητάμε για το γεγονός ότι θέλουμε οι δοκιμές στα ζώα, τα πειράματα στα ζώα να είναι όσο γίνεται πιο περιορισμένα, αλλά τελικά οι αριθμοί αυξάνονται, δεν μειώνονται. Γι' αυτό και χρειάζονται συγκεκριμένοι στόχοι ώστε να επιτευχθεί μείωση των πειραμάτων. Και ένας τρόπος για να το επιτύχουμε αυτό είναι να έχουμε ακριβή στοιχεία. Στοιχεία και να εστιάσουμε την προσοχή μα περισσότερο σε αυτό, γιατί σε πολλούς τομείς ε, δεν χρειάζεται να είμαστε υπερβολικά προστατευτικοί, αλλά πιστεύω πως θα μπορούσαμε να προστατέψουμε πολλά ζώα αν έχουμε καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Και συμφωνώ με την κυρία Μούρκο ότι τα πειράματα σε πρωτογενή, τα, στα πρωτεύοντα θα πρέπει να εξαλειφθούν. Έχει κάνει εξαιρετική έκθεση και μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Και ως ε, πράσινο έχουμε καταθέσει κάποιες ε, τροπολογίες που ελπίζω πως θα μπορέσει να τις υποστηρίξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λεωτάρ. Η κυρία Τζάκσον. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήρθα προετοιμασμένη να πάθω κατάθλιψη μετά όσα θα ακούγα από του συναδέλφου. αλλά η κυρία Φερέρα με χαροποίησε με την έκρηξη κοινή λογική της. Ελπίζω να μην την πειράζει που την επενεί μια Βρετανή συντηρητική, ε, ίσως να τα πω ε, κατηδίαν. Εγώ ήμουν εισηγήτρια στην οδηγία του 1996, ήμουν παιδάκι τότε, κοριτσάκι. Και ήταν η πρώτη έκθεση στην οποία με αφήσαν ελεύθερη. <laughs> Μετά από αυτό Ε δεν με άφησαν πια να κάνω τι ήθελα. Ωστόσο θα πρέπει να κατηγορήσουμε την Επιτροπή εντόνω εδώ και 20 χρόνια, όχι ναι, 23 είναι Καρολίνα. Εν πάση περιπτώσει έχω δει πώς έχει εξελιχθεί αυτή η οδηγία από το 1986 μέχρι σήμερα και από καιρού καιρών εγώ θέτω ερωτήσεις γι' αυτό και η Κομισιόν πολύ, πολύ έχει καθυστερήσει να παρακολουθήσει τι έγινε με αυτή την οδηγία και όταν διαμαρτύρονται όπως διαμαρτύρονται στο προήμιο αυτή τη οδηγία για άνεση εφαρμογή δεν καταλαβαίνω ακριβώ τι εννοούν γιατί λένε, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασία, ενώ άλλα εφαρμόζουν τι μήνυμε απαιτήσει τη οδηγία του 86. Ναι, αυτό συμβαίνει στη ζωή όμω. Αυτό έτσι, έτσι εφαρμόζονται οι οδηγίε του ή άλλω. Δηλαδή, ορισμένα κράτη-μέλη μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο από αυτά που λέει η οδηγία. Αυτά έχει ζωή. Ε, αυτό που δεν μπορούμε να αφήσουμε να γίνει, ορισμένα κρατημένα μην κάνουν απολύτω τίποτα για πολύ καιρό και η Κομισιόν να μην κάνει τίποτα. Χρειάζεται ενημέρωση λοιπόν για αυτά, αλλά η κατάσταση δεν είναι αυτή που λέει η Κομισιόν στο επεξηγηματικό τη σημείωμα. Γιατί θυμάμαι ότι το Λουξεμβούργο για χρόνια ε, ξέφευγε χωρίς να κάνει απολύτω τίποτα για αυτήν την οδηγία. Ελπίζω ότι στη συνέχεια έχει αλλάξει την πρακτική του. Τώρα, σε σχέση και με την Επιτροπή Γεωργίας, αν η Επιτροπή Γεωργίας ε, λαμβάνει υπόψη τις δικές μας τροπολογίες, θα ήταν πραγματικά κάτι το ιστορικό, η ιστορική σημασία και θα πρέπει να το προσέξουμε. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να δίνουμε τόση σημασία στην Επιτροπή Γεωργίας. Τώρα, όσον αφορά τη βιασύνη για κρίση. Εγώ μιλάω αγγλικά, αλλά πολλοί από αυτούς που συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση και διαπραγματεύσει και την κατάθεση τροπολογιών δεν μιλούν αγγλικά, δεν είναι η μητρική τους γλώσσα και αγωνίζονται. Και με εντυπωσιάζει πώς το δέχεσαι αυτό. Αν εγώ δεν ήμουν Βρετανή ή Ιρλανδή θα έκανα μεγάλη φασαρία. Όλοι θα έπρεπε να έχετε αντιρρήσεις, γιατί σας εμποδίζουν να υποβάλλετε τροπολογίες, γιατί πρέπει να βρείτε κάποιον που μιλά αγγλικά για να σας βοηθήσει. Και πιστεύω πως αυτό είναι λάθος. Ο εισηγητή δεν στην Επιτροπή Γεωργία δεν ε, θέτει υποψηφιότητα και πάλι. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο να βιαστούμε για να γίνει η πρώτη ανάγνωση ώστε να το περάσει στη δεύτερη ανάγνωση. Θα έχει φύγει ούτω ή άλλω. Θα βγει στη Βουλή των γυρωτήτων. Για αυτό το θέμα, το είναι ερώτηση που ανέφερε η κυρία Φερέιρα για τη ε, πειράματα σε επιθήκους και πρωτεύοντα. Εγώ πιστεύω πως, για να τα πω έτσι ομά, πιστεύω πως η κυρία Μέρκο, που, την οποία κατά τα άλλα εκτιμώ ιδιαίτερα, εδώ δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να παίξουμε μετά όσα προτείνει στην οδηγία η Κομισιόν για το συνεχιζόμενο ε, επίδομα για την πιθανή χρήση πυθίκων ή πρωτο, πρωτευόντων εκτός από ανθρώπους. Ας μην, ας μην έρθουμε σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό που, τι θα έλεγε η ομάδα της κυρίας Μέρκο και, αν πήγαινε στο γιατρό και της λέγανε ότι δυστυχώς έχουν, βρίσκονται στην πρώτη φάση της ε, ασθένειας Alzheimer και τους έλεγαν ότι υπάρχουν κάποια πολύ καινούργια φάρμακα τα οποία θα μπορούσε να δοκιμάσει αλλά δεν θα το τα σύστηνε. Γιατί, γιατί γνώριζε ότι δεν θέλουν να, ε, γιατί, ε, να γίνονται πειράματα στους πυθίκους και στα πρωτεύοντα ε, ζώα και γι' αυτό δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση. Αυτό ακριβώς λέει η τροπολογία της. Λέει ότι η έρευνα θα πρέπει να προχωρήσει με τη βοήθεια των πρωτευών, των ζώων, των πυθίκων κτλ. Ε, ακόμα και αν υπάρχουν χιλιάδες ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια που περιμένουν σε απελπιστική κατάσταση καινούρια φάρμακα. Φάρμακα τα οποία μόνο σε επιθήκους μπορούν να, να, να δοκιμαστούν. Εγώ είμαι μία εξ αυτών. Ε, όταν ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ε, ε, έγινε διάγνωση με την, για την Πάρκινσον. Τα, χέρια μου ακόμα τρέμουν, αλλά μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω γιατί χρησιμοποιώ ένα φάρμακο το οποίο δοκιμάστηκε σε ζώα, σε πρωτεύοντα ζώα. Και θα συνεχίσω να δουλεύω, να παίζω γκολφ και, και χτυπάω και την μπάλα πολύ ίσια γιατί είμαι πολύ άκαμπτη. Αλλά πραγματικά τι θα λέγατε στους ανθρώπους που είναι στην ίδια θέση για μένα, με μένα. Τι, α, ψηφίσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την γνωμοδότηση που απαγορεύει τη χρήση ζώων ε, στα πειράμα, ε, γιατί μας δείχναν όλες αυτές τις εικόνες για τα, με τα καημένα τα ζωάκια στα εργαστήρια. Μα ποιον θα βάλουμε πρώτα, την ανθρωπότητα ή τα ζώα. Τελικά περί αυτού πρόκειται. Νομίζω πως ε, αυτή η οδηγία την οποία προτείνει η Κομισιόν έχει κάποια λάθη και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε, αλλά εν γέννη έχει βρει καλή ισορροπία σε σχέση με τη συγκεκριμένη πτυχή της χρήσης των πρωτευόντων ζώων και των πυθίκων. Για το θέμα των πυθίκων που λέμε ότι είναι πιο κοντά σε εμά, δεν χρησιμοποιούνται στο ΕΒ και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθόλου. Αλλά αυτό που κάνει η οδηγία είναι να διατηρήσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα σε κάποιο είδο πανδημία που μπορεί να προκύψει, την οποία δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τώρα. Τι θα γινόταν τότε, θα, θα πρέπει να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί αλλιώ εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν. Και εδώ κλείνω αυτό το κομμάτι και τελευταία μου παρατήρηση. Όταν μιλάμε για επιθεωρήσεις, πραγματικά θαυμάζω την ε, ε, πρόταση καμικάζ της κυρίας Μέρκο για τις επιθεωρήσεις, γιατί αντικατοπτρίζει αυτά που προσπαθούσα εγώ να κάνω για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις εν γέννη. Εκείνη θεσπίζει μια επιθεώρηση για αυτό το θέμα. Καλή τύχη, θα δείτε ότι το Συμβούλιο δεν θα τα δεχτεί. Αλλά έχει απόλυτο δίκιο πως αν έχουμε πολύ συγκεκριμένη οδηγία με πολλές λεπτομέρειες που η Κομισιόν είτε δεν μπορεί να εφαρμόσει είτε δεν θέλει να ε, συνεχίσει και να παρακολουθήσει τι κάνουν τα κράτη-μέλη, τότε θα έχουμε δίλημα για το τι να κάνουμε. Θα περιμένουμε τα κράτη-μέλη να μας στείλουν τις εκθέσεις τους που δεν τις στέλνουν, θα στείλουμε επιθεώρηση που δεν έχουμε επιθεωρητές, είτε θα εφεύρουμε μια επιθεώρηση που τα κράτη-μέλη δεν θα μας αφήσουν να φτιάξουμε. Αυτό προσπαθεί να κάνει και τη θαυμάζω γιατί πιστεύω πως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διατηρήσουμε στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής. Αυτά για την ώρα, αλλά σίγουρα θα σας μιλήσω για αυτά ή ίσως και όχι. Για τελική μου παρατήρηση είναι αυτή. Είπε ο κ. Χόπενς όταν τελείωνε ότι προσβλέπει στην περαιτέρω συζήτηση των τροπολογιών. Εγώ από ό,τι κατάλαβα αυτή είναι η τελευταία συζήτηση που θα έχουμε. Δεν θα γίνει καμιά συζήτηση για τις τροπολογίες και αυτό πάλι είναι τελείω λάθος. Και ίσως να μην είμαι σε θέση να είμαι εδώ. Ίσως λοιπόν, να παίξω γκολφ καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζάξον. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Γκροστέτ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο γιατί είμαι εισηγήτρια για την οδηγία αυτή για τα πειράματα στα ζώα στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Και θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα προ την κατεύθυνση των λόγων τη κυρία Τζάξον. Συμφωνώ με του συναδέλφου. Πρέπει να αποφύγουμε τι ε, ε, ε φορτισμένε συναισθηματικά συζητήσει, παρόλο που το 2005 χρησιμοποιήθηκαν 12 εκατομμύρια ζώα ε, για τα πειράματα αυτά. Επί 25 κρατών μελών. Άρα στην πραγματικότητα έχουμε σταθερό ε, αριθμό ζώων, ε, λαμβάνοντα υπόψη ότι αυξάνονται οι δραστηριότητε τη επιστήμη. Άρα η πρώτη οδηγία είχε κάποια αποτελέσματα όσον αφορά την ανάγκη εξέβριση αναλλακτικών μεθόδων. Μία στι 10 ε, το ζώο που χρησιμοποιείται είναι ποντίκι ή αρουραίο και μία στι χίλιε είναι πρωτεύων. Άρα, με βάση όλα αυτά, τώρα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι πράγματι οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να, έτσι ώστε ε, να οδηγηθούν προ εναλλακτικέ λύσει. Αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιπτώσει για τι οποίε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσει. Και η κυρία Φεραίρα το είπε εξάλλου, έτσι. Όταν πρόκειται για ε, έρευνα για το AIDS, για τις ε, νευροεκφυλιστικές ε, ασθένειες, Alzheimer, Parkinson κτλ. Ε, εκεί είναι απαραίτητο να ε, καταφεύγουμε στα πειράματα επί πρωτευόντων. Να σας πω τώρα το εξή. Κοιτάξτε, θα ήθελα να υψίσω την προσοχή των συναδέλφων τη Επιτροπή Περιβάλλοντο στου κινδύνου μια πολιτική ε, που με συστηματικό τρόπο ε, θα οδηγήσει στην έρευνα επί τη δεύτερη γενιά των πρωτευόντων. Στην ουσία, τα ωφέλη από τα πειράματα επί της δεύτερης γενιάς δεν ε, έχουν αποδειχθεί καθόλου. Όσον αφορά την προστασία των ζώων, η ανάπτυξη προγραμμάτων ε, κοινωνικοποίησης αποτελεί ε, βελτίωση των συνθήκων ε, αντιμετώπιση των ζώων αυτών που προορίζονται ε, στην έρευνα. Εξάλλου το συζητάμε με τα επιστημονικά ε, ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης, αν μπορούμε να μιλήσουμε για έρευνα στην Ευρώπη, μας αναφέρουν ότι ε, και για τους ίδιους το βασικό είναι η καλή κατάσταση των ζώων. Γιατί εάν ε, υφίστανται βρίσκονται σε, κάτω από στρες τα ζώα επειδή ακριβώς υποφέρουν, τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα. Άρα πρέπει να καταβάλουν με κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το ζώο του οποίου γίνει το, το πείραμα να μην υποφέρει. Λαμβάνεται λοιπόν υπόψη ευθύ εξ αρχής ε, η, η οδύνη του ζώου και σέβονται όσο το δυνατόν γίνεται την καλή κατάστασή του. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και είναι πολύ σημαντικό, κυρίως αν λάβουμε υπόψη, ότι με τον τρόπο αυτό θα προωθήσουμε την έρευνα στην Ευρώπη ε, γιατί, και τα πειράματα στην Ευρώπη, γιατί εκεί επιβάλλουμε τους δικού μας κανόνες και όσον αφορά το περιβάλλον και την υγεία. Γιατί αν δεν επιτρέπουμε πειράματα με ζώα στην Ευρώπη, τότε αυτά τα πειράματα θα γίνουν, όπως δυστυχώς ήδη γίνονται πολλά σήμερα, σε τρίτες χώρε, στην Ασία για παράδειγμα, χωρί τον παραμικρό έλεγχο από μεριά μα. έλεγχο των συνθήκων κάτω από τις οποίες γίνονται τα πειράματα και ε, την καλή κατάσταση των ζώων που χρησιμοποιούνται. Άρα λοιπόν δεν θα έχουμε πλέον καλά αποτελέσματα. Ας διατηρήσουμε τα πειράματα ε, στην Ευρώπη, γιατί σε αυτή την περίπτωση είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση και ότι ε, η νομοθεσία και οι διατάξεις και τις συγκεκριμένε οδηγίες θα σέβονται. Ε, θα αποτελούν, συγγνώμη, θα αποτελούν το κείμενο σεβασμού και, θα, και ότι ταυτόχρονα θα αποτελεί κείμενο σεβασμού και η καλή κατάσταση των ζώων. Για παράδειγμα, η συστηματική εφαρμογή μιας πολιτικής πειραμάτων στη δεύτερη γενιά θα υποχρεώσει διπλασιασμό των πόρων σε, ε, όσον αφορά ε, την εκτροφή των ζώων και ο, ο παραγωγός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση ε, έναντι και των ανταγωνιστών του στη ΣΥΠΑ ή στην Ιαπωνία. Μην ε, σκοτώνουμε λοιπόν την έρευνα, ας δώσουμε τη δυνατότητα στην έρευνα να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο βεβαίω κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Εξάλλου η πολιτική αυτή θα οδηγήσει στους παραγωγούς σε μαζική ευθανασία των αρσενικών ζώων. Ε, και μην ξεχνάμε ότι στην, εκτροφή των ζώων χρησιμοποιείται ένα αρσενικό για 10 θηλυκά. Ε, ας προσέξουμε λοιπόν Μπορεί να είναι καλέ οι προθέσει μα, αλλά όλα αυτά να στραφούν εναντίον μα. Θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτά τα οποία θα ζητήσουμε και μέσα από την οδηγία αυτή. Τέλο, σα μίλησα για τον κίνδυνο μαζική μετεγκατάσταση των βιομηχανικών ε, δραστηριοτήτων σε χώρε όπω η Κίνα, η Βραζιλία, η Σιγκαπούρη και το γεγονό ότι μπορεί να ε, εκμηδενιστούν τελείω και να ε, φύγουν από το, από το χάρτη ε, ε, εργαστήρια στην Ευρώπη. Και μην ξεχνάμε, όταν συζητάμε με του ερευνητέ, όλοι μα επαναλαμβάνουν ότι δεν έχουν δεν θέλουν να κακομεταχειριστούν τα ζώα που χρησιμοποιούν. Δεν είναι προς το συμφέρον τους. Ε, δεν είναι κάτι τέτοιο στις προθέσεις τους. Το αντίθετο μάλιστα. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας υπενθυμίζω ότι τα πρωτεύοντα ε, ευτυχώς χρησιμοποιούνται μόνο σε επίπεδο 0,1%. Αλλά είναι ε, ουσιαστική συμβολή τους στην, στα, στα ερευνητικά βιοιατρικά σχέδια και πρέπει να στηριχθούμε ε, σε συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία ε, και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ε, την έρευνα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κροστέτ. Ο κύριος Κύριε Πρόεδρε. Είναι μια έντονη συζήτηση, την είχαμε και στο παρελθόν στα πλαίσια της συζήτησης για τα καλλιτικά και την σχετικά επιτυχή προσπάθεια του Κοινοβουλίου να μειωθεί βαθμιαία, αν όχι να καταργηθεί τελείως, ε, ε, να καταργηθούν τελείως ε, οι δοκιμές σε ζώα για τα καλλιντικά. Βέβαια, αυτό δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τα πειράματα για φάρμακα, για ανθρώπους και θεραπείες. Ως προς τα καλλιτικά μπορούσαμε να πούμε ότι αν στο κάτω-κάτω δεν μπορεί να ε, παραχθεί μια νέα ε, γενιά κραγιών χωρίς δοκιμές σε ζώα, είπαμε εντάξει τότε να μην παραχθεί αυτή η σειρά. Μπορούσαμε τότε να πούμε ότι αν δεν εάν δεν θέλουμε να ε, ε, διακινδυνεύσουμε τη μεταγκατάσταση των ε, δοκιμών, θα αλλάξουμε τα, τα πρότυπα της αγοράς. Για τα φάρμακα όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι αν δεν το επιτρέψουμε εδώ πέρα θα μετακασταθούν οι δοκιμές και μπορούμε να απαγορεύσουμε την ε, εισαγωγή των φαρμάκων που θα έχουν επιστοποιηθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλους τους λόγους που ήδη ακούσαμε. Αυτό θα ήταν ε, μια ε, περιφρόνηση των δικαιωμάτων των ασθενών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω όμως ότι όλοι συμφωνήσαμε ότι θέλουμε μείωση. Το reduction είναι ένα από τα τρία R που αναφέραμε, τις τρεις βασικές αρχές ε, στα ε, ε, πειράματα σε ζώα. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Επίσης όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε πιο ισχυρούς κανόνες προστασίας των ζώων, ευζοίας των ζώων για τα ζώα πάνω στα οποία γίνονται δοκιμές οι περισσότερες δοκιμές ακούσαμε ότι γίνονται σε ποντίκια και σε αρουραίους που μπορεί να μην έχουν τόσους υποστηρικτές όσο τα πρωτεύοντα θηλαστικά. Τα πρωτεύοντα θηλαστικά βρίσκονται, συγγενεύουν πολύ στενά με εμά. και για το λόγο αυτό έχουμε συναισθήματα προς τα ζώα αυτά και υπάρχει επιστημονική, και άλλωστε γι' αυτό υπάρχει και η επιστημονική ανάγκη χρήσης τους σε δοκιμές. Είχαμε συζητήσεις ε, και δηλώσεις στο Κοινοβούλιο που κατέστησαν σαφές ότι δεν θέλουμε δοκιμές σε μεγάλα πυθικοειδή. Δεν θέλουμε να συλλαμβάνονται ζώα από τη φύση ε, για τέτοιους σκοπούς. Όπως ακούσαμε, ο αριθμός των μεγάλων ε, πυθίκων που χρησιμοποιείται είναι πάρα πολύ μικρός. Νομίζω ότι τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκαν στη χώρα μου ήταν ε, στη δεκαετία του 1930. Δεν υπάρχει μαζική χρήση μεγάλων πυθικοειδών. Μπορεί κανείς λοιπόν άνετα να πει ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Το θέμα του κυνηγιού των ζώων αυτών ε, είναι επίσης ε, αρκετά σαφές. Πέρα από αυτό όμως χρειαζόμαστε απάντηση σε κάποια ερωτήματα, διότι αν θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό ε, των ζώων στα οποία γίνονται δοκιμές, θα πρέπει να απαντήσουμε στα, στις ερωτήσεις των επιστημόνων, των ερευνητικών επιχειρήσεων κλπ. Μία από τις ερωτήσεις αυτές είναι τι δείχνουν τα στοιχεία ως προς τη δυνατότητα αναπαραγωγής των ε, ζώων δεύτερης, τρίτης γενιάς. Ε, ε, υπάρχουν στοιχεία ότι ίσως μειώνεται η δυνατότητα να παραγωγείς στη δεύτερη, τρίτη γενιά κράτησης των ζώων αυτών. Έχω επισκεφτεί κέντρα που κάνουν δοκιμές σε ζώα. Δύο πράγματα κάνουν εντύπωση και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε οποιαδήποτε ρύθμιση ε, που να ισχύει για όλη την Ευρώπη είναι το κριτήριο της προστασίας των ζώων, ε, της ευρωίας των ζώων, η Φρανσουάς Γκροστέτ μόλις αναφέρθηκε σε αυτό. Έχω δει καλές πρακτικές στο τομέα αυτών και έχω δει και λιγότερο καλές πρακτικές. Επίσης, Καλή πρακτική είναι οι επιχειρήσεις που κάνουν πειράματα να έχουν κάποιον ανεξάρτητο που να αμφισβητεί κάθε που να εξετάζει κάθε αίτημα για ε, δοκιμές σε ζώα. Ίσως κάτι τέτοιο θα ήταν ε, κάτι που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνουμε στα συγκεκριμένα μέτρα. Να υπάρχει αμφισβήτηση, εξέταση του κάθε αιτήματος, της κάθε αίτησης για δοκιμές σε ζώα. Εάν γίνεται αποδεχτή η αίτηση, τότε να μπορούν να προχωρήσουν τα πειράματα. Αλλά έτσι θα έχουμε κάποια εγγύηση, θα παρέχουμε κάποια εγγύηση ότι εννοούμε στα σοβαρά το θέμα της μείωσης των ε, πειραμάτων. Φυσικά θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στις ε, ερευνητικές εταιρείες, ε, στα ε, πανεπιστημιακά ιδρύματα για να βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις στις δοκιμές με ζώα. Αυτή ήταν η αρχή μας στα καλλιτικά. Έπρεπε να ασκούμε συνεχή πίεση και νομίζω ότι τελικά ε, με τα καλλιτικά οι επιχειρήσεις ε, δέχτηκαν ε, την αποδέχθηκαν την πρόκληση και τώρα συνεργάζονται με την Κομισιόν, συνεργάζονται με τους φορείς για να βρουν εναλλακτικέ λύσεις. Και κάτι ακόμα θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν. Υπάρχει ανησυχία σχετικά με την χρήση τις ε, φράσεις ε, ε, παθήσεις που απειλούν τη ζωή ή είναι ιδιαίτερα καταστροφικές. Αυτό νομίζω ότι θα απέκλειε πειράματα για την παχυσαρκία, το ζαχαρόδι διαβήτη και τέτοια. Δεν είμαι βέβαιος εγώ ότι κάτι τέτοιο θα απέκλειε τέτοιες ασθένειες. Δεν είμαι σίγουρος τι σημαίνει ο ορισμός αυτός. Μπορεί ο, καλά, ο διαβήτης, ε, ο σαχαρότης διαβήτης ε, μπορεί ε, να απειλεί τη ζωή ανθρώπων. σίγουρα πάντως είναι κάτι που έχει πολύ σοβαρές συνέπειες. Νομίζω ότι αν υπάρξει ορισμός της έννοιας αυτής θα μπορέσουμε να ανακουφίσουμε κάποιες από τις ανησυχίες και Τέλος, ε, επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα ε, και στην έκθεση και στη συζήτηση που είχαμε, θα πρέπει να ε, διασφαλίσουμε την ενσωμάτωση αναθεωρήσεων στην πρόταση, να γίνονται τακτικές αναθεωρήσεις για να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα, ποιες είναι οι επιπτώσεις, ώστε μελλοντικά κοινοβούλια να μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις ρυθμίσεις ε, σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα και ενδεχόμενα άλλα μέτρα. Ευχαριστώ κύριε Μπόουις, ο Τόμας Ούλμερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για δύσκολη συζήτηση, ε, πόσο μάλλον που δεν γνωρίζουμε τις τροπολογίες των συναδέλφων. Δεν βρίσκω καλή τη διαδικασία τις τροπολογίες δηλαδή να μπορούμε να τις ε, μόνο το να μπορούμε να υποβάλουμε τι τροπολογίε μόνο στα αγγλικά, ε, άλλωστε αποτελεί διάκριση εις βάρος αυτών που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, ούτε βλέπω να είναι απαραίτητο να υιοθετήσουμε μια απόφαση ε, τόσο γρήγορα. 23 χρονών ε, είναι η παλιά οδηγία, ας αντέξει λίγο ακόμα. Ως προς το περιεχόμενο, να πω ότι έχω συζητήσει με δύο μεγάλα γερμανικά πανεπιστήμια συνάντησα τους ε, υπεύθυνους για τα πειράματα και για την ε, προστασία ε, των ζώων. εφαρμόζουν πολύ αυστηρά κριτήρια και πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων. Συμφωνούμε ότι ε, δεν ε, θέλουμε τον πόνο των ζώων, αν και κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί κατά 100% όταν μιλάμε για πειράματα σε ζώα. Ε, κατά κεφαλήν, ε, κατά διάρκεια της ζωής μας, δύο ε, ζώα καταναλώνει, αντιστοιχούν σε κάθε άνθρωπο ε, που πεθαίνουν σε πειράματα. Ε, βέβαια αυτά τα ζώα μπορεί να είναι μικρά, μπορεί να είναι μεγάλα. Κάποια ζωικά είδη λόγω της στενής συγγένειας με τους ανθρώπους τους ε, προκαλούν ιδιαίτερες ανησυχίες. Η Λίγα όμως είναι τα πειράματα ε, στα οποία είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν τέτοια ζώα. Δύο τέτοια μπορώ να σας ε, αναφέρω. Το ένα είναι η ε, παραγωγή εμβολίων για την υπατήτηδα, για παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας ε, χωρίς τις δοκιμές σε πρωτεύοντα θηλαστικά. Επίσης, απαραίτητα είναι τα ζώα αυτά για τις χειρουργικές έρευνες. θα πρέπει να ε, θέσουμε συγκεκριμένα όρια ε, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των ε, πειραμάτων σε ζώα δεν είναι ιδιαίτερα θετικά. Ε, θα πρέπει κάποιες επιτυχές ε, να αποτελέσουν ε, αντικείμενο της διαδικασίας της επιτροπολογίας, κάποια, κάποιες πτυχές τις οποίες δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε εμείς. εγώ βλέπω για παράδειγμα ένα πρόβλημα σχετικά με την πιστοποίηση για τους ανθρώπους που κάνουν πειράματα σε ζώα. Η πιστοποίηση αυτή περιορίζεται σε πενταετία, αυτό βρίσκω ότι είναι προβληματικό. Άλλωστε, εάν ε, μεταφερθούν τα πειράματα αυτά εκτός Ευρώπης, τότε δεν έχουμε πετύχει τίποτα ούτε για την προστασία των ζώων, ούτε για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ούλμερ. Η κυρία Καρολάιν Λούκας έχει τώρα το λόγο. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μέρκο για την πολύ καλή έκθεσή της. Λυπάμαι που άργησα και έχασα την εισαγωγή της. Ε, Άκουσα τις παρατηρήσεις της πατριώτησάς μου, της κυρίας Τζάξον και θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Ε, συμμερίζομαι τις ανησυχίες της σχετικά με το γεγονός ότι οι ε, τροπολογίες δεν θα είναι διαθέσιμες σε άλλες γλώσσες. Αυτό σίγουρα είναι ε, δυσάρεστο, αλλά γενικά πιστεύω ότι θα πρέπει να αμφισβητήσουμε αυτήν την ε, πολύ γρήγορη διαδικασία που μας έχει επιβληθεί. Χρόνια περιμένουμε την επανεξέταση της ε, πρότασης. Ο Νίλ Πάρης θα αποχωρήσει από το Κοινοβούλιο για την ε, Βουλή των ε, ε, κοινοτήτων στην Βρετανία. Χαίρομαι που τελικά επιτέλους η Κομισιόν υπέβαλε την πρόταση αυτή. Το άλλο θέμα που θα ήθελα να σχολιάσω ε, από αυτά που είπε η κυρία Τζάξον ε, και νομίζω ότι είναι λεπτό θέμα για όλους μας είναι ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε από την αντίθεση ανάμεσα στην προστασία της ε, ανθρώπινης υγείας και την προστασία των ζώων. Δεν είναι πάντα οι δοκιμές σε ζώα ο καλύτερος τρόπος να διαπιστωθεί το αποτέλεσμα σε ανθρώπους. Κάποια εργαστήρια στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, κάνανε πειράματα σε ανθρώπους που είχαν γίνει ήδη σε ζώα. Τα αποτελέσματα δεν ήταν πολύ καλά. Οι άνθρωποι σχεδόν πέθαν, πέθαναν. Ε, επίσης ε, έχουμε δει αρνητικά αποτελέσματα σε ζώα και θετικά αποτελέσματα σε ανθρώπους. Αν κοιτάξουμε τις δοκιμές σε ζώα πιο προσεκτικά θα δούμε ότι πολλά, πολλές δοκιμές δεν δίνουν σαφή αποτελέσματα. Ε, πολλά, πολλές δοκιμές ε, έχουν ε, αποτέλεσμα 50-50 ε, κατά την επανάληψη των δοκιμών. δηλαδή 50% είναι η πιθανότητα να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα αν επαναλάβουμε κάποια δοκιμή, το οποίο συμβαίνει και όταν ρίχνουμε ένα νόμισμα κοροναγράμματα. Νομίζω ότι είναι δυνατή η πρόωθηση εναλλακτικών λύσεων ε, που θα είναι καλές και για τα ζώα και για τους ανθρώπους ε, και υπάρχουν πολλές εναλλακτικέ λύσεις. Θα πρέπει όμως να επιταχύνουμε την έρευνα των διαδικασιών αυτών, την πιστοποίησή τους και τη διάθεσή τους ε, στην αγορά. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει να κάνει η έκθεση της κυρίας Μέρκο. Ε, εντύπωση μου έκανε αυτό που είπε ο κύριος Μπόης, ότι θα πρέπει να πιέσουμε όλους τους παράγοντες ε, στη διαδικασία αυτή για να ε, βρεθούν εναλλακτικέ λύσεις. Μου φαίνεται όμως ότι όπως έχει η πρόταση της Επιτροπής αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αρκετό κίνητρο ή επαρκής πίεση για να ε, ε, βρεθούν αυτές οι εναλλακτικέ μέθοδοι. Νομίζω θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Ε, εγώ θα υποβάλω τροπολογία ε, ώστε να δημιουργηθούν όχι μόνο εθνικά κέντρα αριστείας αλλά και ένα ευρωπαϊκό κέντρο συντονισμού για εναλλακτικέ μεθόδους. Από τα 12 εκατομμύρια ζώα που χρησιμοποιούν το 2005 για επιστημονικούς ε, σκοπούς, το 80 ε, ή 90% ε, χρησιμοποιήθηκαν για βιοφαρμακευτικές και κτηνιατρικές έρευνες. Οι διαδικασίες αυτές ε, δεν καλύπτονται από την ΕΚΦΑΜ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο ε, για την ε, επιστοποίηση των εναλλακτικών μεθόδων. Πιστεύω θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις τρεις αρχές, τα τρία ρο που λέμε, την μείωση, την αντικατάσταση και την εξέλιξη των μεθόδων σε όλες τις διαδικασίες, όχι μόνο σε αυτές που καλύπτονται από την ΕΚΦΑΜ. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη χρήση εναλλακτικών λύσεων ε, και θα πρέπει να συντονίσουμε τις έρευνες που γίνονται σε εθνικό επίπεδο στις διάφορες χώρες θα πρέπει να εξετάσουμε ε, τις ε, διαδικασίες πιστοποίησης που γίνονται από τα εθνικά κέντρα. Θα πρέπει να γίνουν διαβολεύσεις με ενδιαφερομένους ε, για να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή. Κάτι που επιθυμούμε όλοι μας, ώστε να έχουμε πιστοποιημένες εναλλακτικέ λύσεις οι οποίες να διατεθούν στην αγορά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μέρκο για την έκθεσή της. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ καλό υλικό εδώ πέρα, το οποίο θα έχει καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τέλος η κυρία Ντάγμα Ροκμένετ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μάλλον δεν θα έπρεπε να μιλάω. Αλλά δεν αντέχω. Ε, αν και η φωνή μου δεν πάει πολύ καλά. Γνωρίζετε ότι εδώ και 15 χρόνια ή περισσότερο ακόμα αγωνίζομαι για την απαγόρευση των πειραμάτων σε ζώα για τα καλλιτικά. Αγωνίστηκα διότι με την υποστήριξή σας ήθελα να πω ότι το προϊόν έχει σημασία για ποιο προϊόν γίνονται δοκιμές σε ζώα. Όλα αυτά τα χρόνια έλεγα όμως ότι δεν αγγίζω καν το θέμα των δοκιμών σε ζώα για φάρμακα. Και δεν το κάνω αυτό διότι δεν θα ήθελα να βρεθώ στη θέση να συζητήσουμε για ποιες ασθένειες επιτρέπεται να γίνουν πειράματα σε ζώα και ποιες είναι οι ασθένειες που δεν είναι αρκετά σοβαρές ώστε να γίνονται πειράματα σε ζώα. Σήμερα στη συζήτηση το ακούσαμε αυτό άλλωστε. Δεν θέλω να συζητήσω τι απειλεί τη ζωή ή απλά επιβαρύνει, ε, επιδεινώνει την ποιότητα ζωής κάποιου. Δεν θα βγω εγώ μπροστά σε μια οργάνωση ασθενών και να πω ότι τα παιδιά σας ε, τα παιδιά σας υποφέρουν ε, από ε, χρόνια πάθηση, αλλά εμείς θα σταματήσουμε τα πειράματα σε ζώα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνονται πειράματα σε ζώα χωρίς οποιαδήποτε, χωρίς περιορισμό και χωρίς τις τρεις βασικές αρχές, χωρίς ελέγχους. Συμμερίζομαι τη θέση της κυρίας Τζάξον. Πιστεύω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούμε να έχουμε επιθεωρήσεις. Πολύ ωραίο αυτό, αλλά είναι και αφελές. Δεν, δεν το πετυχαίνουμε αυτό ούτε στον τομέα των τροφίμων. Από τότε με την σπογκώδη εγκεφαλοπάθεια δεν έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε, ε, να κάνουμε τέτοιους ελέγχους. Ούτε σε άλλους τους τομείς θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τα εργαστήρια. Ωραία προσπάθεια, αλλά κανένα κράτος μέλος δεν πρόκειται να δώσει πόρους για κάτι τέτοιο. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Κυρία Μούρκο, πιστεύω έχει μια πολύ καλή προσέγγιση. Αλλά εγώ βρίσκω υπερβολικές κάποιες από τις προτάσεις της. Και το λέω αυτό ζυγίζοντας τα ωφέλη και τις ασθένειες που θέλουμε να θεραπεύσουμε. Εάν μπορούμε in vitro να θεραπεύσουμε τις ε, ασθένειες αυτές, τότε να το κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα απαιτήσει πολύ χρόνο. Ε, θέλουμε να χρησιμοποιούμε όσο γίνεται λιγότερα ζώα και ε, τα ζώα αυτά να υποφέρουν όσο γίνεται λιγότερο. Το θέμα δεν είναι αν θα έχουμε τις τροπολογίες μόνο στα αγγλικά. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε όλες τις τροπολογίες και στα αγγλικά. Λυπάμαι. Ιδιαίτερα που η πρόταση αυτή της Κομισιόν υπάρχει από τον Νοέμβριο και που δεν τη συζητήσαμε νωρίτερα. όποιος ενδιαφερόταν για το θέμα μπορούσε να το εξετάσει εγκαίρως. Κρίμα που δεν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε. Και ε, αφήνω τελείως ε, κατά μέρος το ε, πρόβλημα της σύγκρουσης των συμφερόντων, το, αν, το ποια επιτροπή θα έπρεπε να αναλάβει το θέμα αυτό. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο Ευρωπαϊκό Κέντρο. Αγωνίστηκα χρόνια για την ύπαρξη του ΕΚΦΑΜ και γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα που έχει το κέντρο αυτό. Αγωνίζεται για να έχει αρκετά χρήματα, να έχει επαρκή τεχνογνωσία και να βρει την ισορροπία ανάμεσα στο να βρει ε, εναλλακτικές λύσεις ε, ή το να πιστοποιητική εναλλακτικές λύσεις. Τώρα το να δημιουργήσουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό κέντρο βρίσκω την Είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να τα χαλάσουμε όλα. Πρέπει να ενισχύσουμε το ΕΚΦΑΜ. Δεν έχω πρόβλημα ε, με το μέρος στην Ιταλία που θα βρίσκεται το κέντρο. Ε, είναι πολύ ωραίο. Αλλά ε, έχουμε ήδη τσακωθεί μεταξύ μας για το πόσα χρήματα θα πρέπει να έχει ο προϋπολογισμός της ΕΚΦΑΜ. Ίσως θα ήταν αυτό μια αφορμή να κάνουμε κάπως καλύτερα τα πράγματα. Θέλουμε να πετύχουμε λιγότερα πειράματα σε ζώα για τα φάρμακα. Η μόνη εναλλακτική λύση είναι να προωθήσουμε ε, εργαστηριακές ε, δοκιμές, εναλλακτικές μεθόδους. Ήδη αν πετύχουμε κάτι τέτοιο κατά 70% θα είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα. Για κάτι τέτοιο απαιτούνται οι προσπάθειες του σχετικού ε, τομέα, της φαρμακοβιομηχανίας δηλαδή, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ροτπέραντ. Εύχομαι η φωνή σας ε, να επανέλθει σύντομα. Να ξεκουραστείτε. Έτσι κλείνουμε το κατάλογο των ομιλητών. Θα ε, απευθυνθώ τώρα στην εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν, την κυρία Σχόνμακερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την Επιτροπή για την ε, τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπως είπε ο κύριος Μπόης, ε, ε, και ιδιαίτερα πλούσια συζήτηση. 9,5 σελίδες σημειώσεις κράτησα και να προσπαθήσω να τοποθετηθώ σε όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και βεβαίως δεν μπορώ να καλύψω στις λεπτομέρειες τα πάντα. Θα ήθελα βεβαίως να πω αυτής εξ ότι η συζήτηση ε, αντικατοπτρίζει πολύ πιστά, αν θέλετε, και τη συζήτηση με τους εμπλεκόμενου και με του ενδιαφερόμενους, μετά ε, ε, τη συζήτηση με βάση την πρόταση τη Επιτροπή, αλλά και εντός τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η συζήτηση αυτή, όπως ήδη τόνισαν πολλοί προραλίσσαντε, προσπαθεί να ε, υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στα δύο συμφέροντα, τα οποία δεν είναι εμφυλεγόμενα, αλλά πρέπει βεβαίω να συμφιληθούν σε μια οδηγία. Το βασικό μας ε, ενδιαφέρον είναι η ε, σημαντική ε, αύξηση της ευζοίας, αλλά με έναν τρόπο που να μην καταστρέφει ή να παρεμποδίζει την έρευνα και να μην έχει αρνητικά, αρνητικές επιπτώσεις και στη φαρμακοβιομηχανία. Και βεβαίως ε, δεν θέλουμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου ε, ε, οι φαρμακοβιομηχανίες και οι ερευνητές θα θεωρήσουν ότι είναι πιο εύκολο να μετεγκατασταθούν εκτός Ευρώπης, διότι εκεί η έρευνα γίνεται με πολύ χαμηλότερα πρότυπα και, και διατάξεις και ε, διαφεύγει από τον έλεγχό μας. Το θέμα είναι πώς θα υπάρξει η ισορροπία αυτή. Και θα ήθελα να τονίσω ε, στην απάντησή μου ότι εμείς ε, εδώ ε, συμπεριλάβαμε ορισμένα στοιχεία για να είμαστε σίγουροι ότι έχει αυξηθεί η καλή κατάσταση των ζώων. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην υποχρεωτική άδεια για όλα τα σχέδια τα οποία ε, λαμβάνουν χώρα και την ε, ε, ηθική αξιολόγηση όλων των σχεδίων και την αξιολόγηση από άποψη ευεντολογία. Αλλά βεβαίω και αυτό βεβαίω αποτελεί βάρο για τα ερευνητικά ιδρύματα και για τη βιομηχανία και προσπαθήσαμε εδώ να ακολουθήσουν μια ρεαλιστική προσέγγιση. Και, και είπαμε ότι ορισμένες ε, διατάξεις ε, ε, θα πρέπει να διευκολύνουν τις ομαδικές άδειες, αν θέλετε για παράδειγμα, ή την περίπτωση, εάν μέσα σε 30 μέρες δεν έχει απαντήσει η διοίκηση, να θεωρήσουν ότι έχει δοθεί η άδεια καταρχήν. Επίσης, η αύξηση διαφάνειας, πολύ σημαντική για την ε, αύξηση της συμμόρφωσης και εδώ περιέχονται πολλές διατάξεις προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ε, παραπέμπω ιδιαίτερα ε, στις συνόψεις των μη τεχνικών σχεδίων, αλλά και στην εκ των υστέρων αξιολόγηση. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, Πέραν αυτών των γενικών σχολείων, θα ήθελα να τοποθετηθώ και να απαντήσω σε ορισμένα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν. Θα προσπαθήσω να καλύψω στον μετώπιση περισσότερε ερωτήσει σε κάποια λογικά χρονικά πλαίσια και ε, είμαι έτοιμη για περαιτέρω συζήτηση, αν το επιθυμείτε. Πρώτα απ' όλα, έγιναν διάφορα σχόλια προ διάφορε κατευθύνσει όσον αφορά την απαγόρευση τη χρήση των μεγάλων πυθικοειδών και επίση ε, όσον αφορά τη σταδιακή απαγόρευση ε, τη χρήση των μη ανθρωπίνων πρωτευόντων. Κοιτάξτε, ακολουθήσαμε την πρώτη οδό, αλλά δεν θεωρήσαμε ότι είναι λογικό, και αυτό το είπαν και πολλοί ομιλητέ σήμερα το απόγευμα, ότι είναι λογικό να κλείσουμε την πόρτα για πάντα σε, ε, σε, ε, σε κάθε έρευνα προ την κατεύθυνση αυτή. Δεν θέλουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου τελικά θα αναγκαστούμε να θυσιάσουμε την ανθρώπινη ζωή, επειδή δέσαμε τα χέρια μα μόνοι μα και ε, δεν θα επιτρέπεται ε, οποιοδήποτε συνθήκη κάτω από οποιοδήποτε συνθήκε να, ε, να γίνουν πειράματα στα μεγάλα πυθικοειδή. Έχουμε όμω ιερήτερη διασφάλιση. Όπου λέμε ότι αν γίνεται τέτοια έρευνα θα πρέπει να γίνεται κάτω από εξαιρετικέ συνθήκε που περιγράφονται στην οδηγία και απαιτείται άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η άδεια αυτή θα δοθεί μόνο ε, εάν έχει, γίνει, ε, έχει περάσει από τη διαδικασία της επιτροπολογίας με το Κοινοβούλιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δικλείδες ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των ε, ζώων αυτών. Επίσης, πολλοί είπαν ότι θα πρέπει να ε, απαγορευτεί, ε, η, απαγορευτούν τα πειράματα σε μία ανθρώπινα πρωτεύοντα. Συμφωνούμε. έχουμε λάβει την άποψη όλων των επιστημονικών επιτροπών και φαίνεται ότι δεν είναι ακόμα εφικτό να δώσουμε συγκεκριμένε προθεσμίες. Γνωρίζουμε ότι θα συνεχίσει να είναι απαραίτητη η έρευνα αυτή για λίγο και πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου όλο και λιγότερο ε, καταφεύγει η επιστήμη σε αυτά τα πειράματα. Προσπαθούμε πάντα να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογή τη έρευνα αυτή και ε, τοποθετήθηκε ο κ. Μπόβη στο θέμα αυτό και μα ε, ρώτησε ε, για το ποιε είναι αυτές οι συνθήκε που απειλούν τη ζωή ή αποδυναμώνουν την ε, υγεία του ανθρώπου. Οι όροι αυτοί ε, δεν ορίζονται συγκεκριμένη νομοθεσία, αλλά ορίζονται αλλού στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και βεβαίω περιγράφουμε κάπω τα πράγματα στις αιτιολογικές σκέψεις. Εκεί ορίζουμε ε, αυτές τις ε, καταστάσεις ως καταστάσεις ε, που έχουν σημαντική επίπτωση στην καθημερινή λειτουργία του και δραστηριότητα του ασθενού. Και νομίζουμε ότι αυτοί, αυτές οι περιγραφές είναι αρκετά αυστηρές, αλλά αφήνουν το απαραίτητο περιθώριο λιγμών, το οποίο χρειάζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Χρειαζόμαστε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όσον αφορά του ελέγχου τώρα, έγιναν διάφορες ερωτήσεις η οδηγία προβλέπει τη σημαντική ενίσχυση του συστήματος ελέγχων έναντι τη υφιστάμενη κατάσταση. Σήμερα μιλάμε για περιοδικούς ελέγχους που καλύπτουν τα πάντα, κάθε 5 χρόνια, κάθε 10 χρόνια. Ενώ η οδηγία προβλέπει οι εθνικές διοικήσεις να προβαίνουν σε ελέγχους δύο φορές το χρόνο. Τώρα, ακούσαμε την εισηγήτρια για κάποιου άλλου να υποστηρίζει την άποψη ότι όλα αυτά δεν αρκούν. Ε, ναι, τότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα για ε, έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα ελέγχει, αν θέλει, του εθνικού ε, ελεκτέ, Αλλά και εγώ, όπω και η κυρία Τζάξον, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Και α δούμε πώ ε, θα λειτουργήσουν τα πράγματα. Έχουμε την πρόταση για ενίσχυση των ελέγχων. Εάν ε, θεωρήσουμε ότι είναι απαραίτητο, τότε να κατεβάσουμε και το βαρύ πυροβολικό όσον αφορά του ελέγχου, που ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν σε αυτήν την περίπτωση. Τώρα, έγιναν κάποια, κάποια άλλα σχόλια όσον αφορά τα κριτήρια για την ταξινόμηση. Δεν θέλω να επισέλθω σε τέτοιε λεπτομέρειε. Απλά και μόνο να σα πω ότι ναι, βεβαίω, ε, έχουμε εδώ ένα σύστημα ταξινόμηση με διαφορετικέ υποχρεώσει που συνδέονται με κάθε ε, ταξινόμηση. Το σύστημα ταξινόμηση στην οδηγία δεν ε, περιγράφεται με ακρίβεια, αλλά να πω το εξή, ότι στα πλαίσια τη ερευνητική κοινότητα Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπάρχει ε, συνένεση όσον αφορά το τι αφορά ήπια ή σοβαρή διαδικασία. Υπάρχουν βεβαίω κάποιε φαιέ ζώνε που θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Γι' αυτό όμω έχει ξεκινήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπουμε μέχρι να αρχίσει να τίθεται σε ισχύ η οδηγία τότε εμείς θα έχουμε ε, πρόταση μέσω της επιτροπολογίας για να ορίσουμε περαιτέρω αυτά τα κριτήρια. Τώρα, τι άλλο θέλω να πω. Έγιναν διάφορα σχόλια ε, που, ε, όσον αφορά την ανάγκη ανταλλαγή στοιχείων. Βεβαίω, αυτό είναι μια τάση που ήδη διαφαίνεται στην ε, νομοθεσία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράδειγμα, παρεστοκτόνα. Πιστεύουμε ότι οι διατάξεις αυτές ε, βρίσκονται ε, με καλύτερο τρόπο στις τομιακές νομοθεσίες. Ναι, καταλαβαίνω, Πρόεδρε, δεν έχω αρκετό χρόνο. Αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια για το θέμα τη μετακίνηση προ τη γενιά F2. Έγιναν σχόλια. Ορισμένοι υποστηρίζουν την πρόταση τη επιτροπή αλλά ορισμένοι εκφράζουν ανησυχίε. Στο τι θα συνεπάγεται κάτι τέτοιο για την ερευνητική κοινότητα. Η ιδέα τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής είναι η εξή. ή μάλλον να το πω διαφορετικά, λαμβάνει υπόψη τα διάφορα στοιχεία τα οποία ακούστηκαν εδώ και προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, δίνοντας αυτήν μετακίνηση προ δεύτερη γενιά ή ακόμα και υψηλότερα, αλλά ταυτόχρονα προβλέπουμε υποβολή έκθεση από τα κράτη-μέλη όσον αφορά την προέλευση των μη ανθρωπο, ανθρώπινων προβλητευόντων και επίσης προβλέπουμε αξιολόγηση των επιπτώσεων και όσον αφορά την κατάσταση των ζώων και τις οικονομικές επιπτώσεις. Θα υπάρξει δυνατότητα λοιπόν αθεώρηση των διατάξεων της οδηγίας εάν προκύψει ανάγκη. Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά τις προθεσμίες για σταδιακή αντιμετώπιση ε, προήλθαν ε, από ε, Επιστημονική Επιτροπή συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι και εκπρόσωποι της βιομηχανίας και οι προθεσμίες για σταδιακή μείωση λαμβάνουν υπόψη το χρόνο εκτροφής του ζώου καθώς επίσης τη διαθεσιμότητα ορισμένων ζώων τη κατηγορίας F1, δηλαδή πρώτης γενιάς ζώα σε εχμαλωσία. Νομίζω ότι θα ήθελα να σταμα... μάλλον πρέπει να σταματήσω εδώ. Σημειώσαμε την... Ε, το γεγονός ότι για άλλη μια φορά απευθύνεται έκκληση για εργασία προς την κατεύθυνση των ελεκτικών μεθόδων, έτσι ώστε και να ενισχυθεί και το γεγονός ότι ζητάτε να ενισχυθεί ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν ορισμένα μέτρα που ήδη αναφέρονται στην οδηγία και όπου προβλέπουν τη δημιουργία ε, εθνικών εργαστηρίων αναφοράς που θα τα συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βεβαίω, όταν μιλάμε για, για συντονισμό από την Επιτροπή βεβαίω καλύπτουμε ε, όλες τις πιθανότητες στις οποίες αναφερθήκατε και εσείς. Και τέλος να πω το εξής. Προς το τέλος Δεκεμβρίου η Επιτροπή ε, τοποθετήθηκε και υπέβαλε έκθεση όσον αφορά τι διάφορε δεσμεύσει που αναλάβαμε ενώπιον του Κοινοβουλίου. Ψήφισμα ε, Μαΐου για, την, για τις μεθόδους ε, δοκιμών και και εδώ λάβαμε συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένη οδηγία και για να ενισχυθεί η δαφάνεια και κυρίω να επιταχυθεί η διαδικασία επαλήθευση. Κύριε Πρόεδρε, συνειδητοποιώ ότι δεν έχω απαντήσει σε πολλέ ερωτήσει, πολύ συγκεκριμένε. Δεν νομίζω ότι ε, μπορώ να ε, ε, κρατήσω το ενδιαφέρον σα για περισσότερο χρονικό διάστημα. Πολύ ευχαρίστω όμω αν κάποιο θέλει μια συγκεκριμένη διασαφήνιση. Ευχαριστώ. Mevrouw Jackson heeft om het woord gevraagd. Mevrouw Jackson. Σας ευχαριστώ κυρία Τζάκσον να ζητήσω το λόγο. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να κάνω άλλη μία συναισθηματική επίπεδη για το θέμα του χρόνου. Οι εκπρόσωποι της Κομισιόν μπορούν να μας πούν ποια είναι τα προγράμματα της Προεδρίας του Συμβουλίου πότε προγραμματίζουν να υιοθετήσουν την πρώτη ανάγνωση και ελπίζουν να υπάρξει συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση, πράγμα το οποίο θα ήταν πολύ ανεπιθύμητο για μας. Ποιο, είναι το χρονοδιάγραμμα του Συμβουλίου. Κοιτούσα γύρω μου να δω πως υπάρχουν εκπρόσωποι του Συμβουλίου, αλλά δεν είδα κανέναν. Δεν γνωρίζω, πρέπει να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα αρχίσει τη συζήτηση στο Συμβούλιο. Νομίζω αυτή τη βδομάδα θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις ή την επόμενη. Με μισό λεπτό. Δύο συνεδριάσεις προβλέπονται για την αρμόδια ομάδα εργασία που είναι και υποομάδα του Συμβουλίου για τη Γεωργία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε σαφεί ενδείξει από την Προεδρία για ποιο βαθμό προτεραιότητας θέλουν να δώσουν αυτό το θέμα και δεν νομίζω πως θα στοχεύουν σε συμφωνία πρώτης ανάγνωσης, τότε γιατί βιαζόμαστε, Πρόεδρε, εμείς. Where's Εμείς βιαζόμαστε, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε την επιρροή μας. Θέλουμε να επηρεάσουμε τη συζήτηση στην Επιτροπή Γεωργίας. Γι' αυτό το λόγο βιαζόμαστε. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Μα ε, ούτω ή άλλω ξέρουμε πω δεν πρόκειται να μα επιλάβουν υπόψη. Αλλά ε, πιστευτείτε με, θα, θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να λάβουν υπόψη τα σχόλιά μα. Ευχαριστώ, κυρία Μπουρκ, Μέρκο. Θέλετε να κλείσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ όλου του ομιλητέ. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του συναδέλφου John Bowies ως σλόγγαν, ως σύνθημα. Να πιέσουμε τη βιομηχανία, τον κλάδο μάλλον, ώστε να βρεθούν εναλλακτικέ για τις δοκιμές στα ζώα. Το θέμα είναι πώς θα το καταφέρουμε αυτό, πώς θα συνεχίσουμε να τους πιέζουμε. Η πλειοψηφία της σημερινής συζήτησης θα έλεγα πως μπορεί όπως ακούσαμε και αρκετές φορές με το, στη σημερινή συζήτηση και από την ερευνητική κοινότητα, ε, καταρχήν ο κλάδος ο ίδιος προσπαθεί προσπαθεί να μειώσει τα πειράματα σε ζώα ή να τα αντικαταστήσει λόγω του κόστους. Το κόστος των εναλλακτικών λύσεων είναι χαμηλότερο από ό,τι δοκιμές σε ζώα. Οπότε δεν χρειάζονται ιδιαίτερα κίνητρα νομοθετικά γιατί η επιστήμη ίδια δουλεύει για την ε, μείωση, την τελειοποίηση και την αντικατάσταση. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή είναι μια λάθος οπτική γωνία. Όλοι συμφωνούμε πως χρειάζομαστε αποτελέσματα, νέα φάρμακα, νέα ε, αποτελέσματα επίσης στην έρευνα, ιδιαίτερα στην ιατρική. Αλλά διαφωνούμε για την μέθοδο που, μέσω της οποίας θα φτάσουμε σε αυτό το σκοπό. Αν και αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλει ιδιαίτερα η φαρμακοβιομηχανία, από το 1986 έχουμε μάθει από άλλους τομείς, ιδιαίτερα από τα τομέα των καλλιτικών, πως η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η εμπλοκή της έχει παίξει ρόλο επιταχυντή όσον αφορά τον περιορισμό των πειραμάτων σε ζώα. Δηλαδή λειτουργούν οι στόχοι. Έχουμε τώρα κάποιες ιδέες για το πώς όλα αυτά θα μετατραπούν σε πράξη και πώς όλα αυτά θα μετατραπούν σε πράξη σε έναν άλλο τομέα. Το θέμα είναι λοιπόν πως ε, ορισμένες φορές τα πειράματα σε πρωτεύοντα είναι απαραίτητα. και ότι το ότι γεγονός ότι αυτά τα είδη κινδυνεύουν δεν είναι τόσο σημαντικό όσο είναι η ε, ανέβρεση νέων φαρμάκων ορισμένες φορές για σημαντικές ασθένειες. Τώρα όλοι μιλάμε για την ε, εξέλιξη. Έχουμε αποτελέσματα και στην εξελικτική ανθρωπολογία που δείχνουν πως και τα πρωτεύοντα βοηθούν στην εξέλιξη. Μαθαίνουμε πολλά περισσότερα για την κοινωνική συμπεριφορά των ε, πρωτευόντων ζώων, ε, για την συνείδησή τους, ε, για τις ομοιότητες και φυσικά και νιώθουν πόνο και υποφέρουν στην απομόνωση. Αυτή είναι μια οπτική γωνία που δεν υπογραμμίστηκε αρκετά σήμερα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που περιορίζουν τις ιατρικές έρευνες. Για παράδειγμα, πολύ καλύτερα φάρμακα θα έχουμε όταν επιτραπείουν οι έρευνες στα βλαστικά κύτταρα. Γιατί δεν το επιτρέπουμε, γιατί είναι ηθικό το ζήτημα. Είναι παράλογο, μα είναι ηθικό. Γιατί ως ανθρωπότητα έχουμε αναπτύξει κάποιους κανόνες και δεν θέλουμε να τους παραβούμε. Δεν είναι ακριβώ το ίδιο, αλλά προσπαθώ κάπως να εξηγήσω από φιλοσοφικής άποψης την άποψή μου. Έχουμε προχωρήσει πολύ από τότε που ξεκίνησαν τα πειράματα σε ζώα για την ε, νόσο του Αλσχάιμερ. Τα ζώα αυτά ωστόσο υποφέρουν και οι μέθοδοι στις οποίες χρησιμοποιούνται τα πρωτεύοντα ζώα πραγματικά είναι ε, φρικτές πολλές φορές. Um, uh, this is ethical angle, but there are other angles and uh, Μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλα πράγματα όπως ότι ότι υπάρχουν δύο βασικοί τομείς ε, δοκιμών. Το ένας είναι ο ρυθμιστικός και η, χρήση, μεγαλύτερη χρήση γίνεται των πρωτοϊβόντων ε, στα εργαστήρια και από την άλλη πλευρά έχουμε γενικές δοκιμές για πειράματα για νέα φάρμακα. Ο τρίτος τομέας είναι τα πειράματα στην ε, βιοπικιλότητα και ιδιαίτερα για νευρολογικές έρευνες. Οι μελέτες αυτές, από όσο γνωρίζουμε, προκαλούν φρικτό πόνο και μπορούν να σημαίνουν την ε, φύτευση ηλεκτρονικών ε, ε, μπίπερ ή τσίπς ε, μέσα στο σώμα των ζώων και δεν ξέρουμε αν όλα αυτά θα φέρουν ωφέλη για την ανθρώπινη υγεία. Να τονίσω πως έχουμε σύγχρονες μεθόδους ανείχνευσης, scanning, για να βλέπουμε εικόνες του ανθρώπινου εγκεφάλου που μας δίνουν ε, κατανόηση άνευ προηγουμένου για τις ψυχικές ασθένειες, τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, τα προβλήματα κοής, όρασης, ομιλίας κτλ. Όλα αυτά δίνουν στοιχεία άμεσης σε σχέσεις με τους ασθενείς που μπορούν Μπορεί να του ζητηθεί, να ερωτηθούν για το πώς αισθάνονται εκείνη τη στιγμή. Το 2008 μια συνεδρίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε όπου παρουσιάστηκε σύγκριση στοιχείων από τις μελέτες κάνει σε ανθρώπους και τα ηλεκτρόδια τα οποία ε, είχαν φυτευτεί στην καρδιά των πυθίκων. Ακριβώς το ίδιο επίπεδο στοιχείων ε, πετύχαμε και το πρώτο ήταν ε, από ανθρώπους. Γιατί λοιπόν συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό στα ζώα αφού δεν το χρειαζόμαστε πια. Ιδού ποια είναι, ποιο είναι το θέμα. Και να τονίσω ότι τα πρωτεύοντα συνήθως έρχονται στο τέλος της στρατηγικής δοκιμών μαζί με τους σκύλους. Πληρούν τις απαιτήσεις δοκιμών σε ένα δεύτερο θηλαστικό εκτός από τα τροκτικά. Και οι πίθηκοι χρησιμοποιούνται στο τέλος του πειράματος, ενώ χιλιάδες άλλα μικρά ζώα έχουν ήδη πεθάνει για το ίδιο προϊόν. Η Κάρολαϊν Λούκας ανέφερε το πείραμα στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο ένα φάρμα, το TG, φάρμακο, το TGN 1412, που προκάλεσε φρικτές και ίσως ε, και θανατηφόρα ή μόνιμες παρενέργειες σε ανθρώπους εθελοντές. Αυτό δοκιμάστηκε αρχικά σε εργαστήρια 500 φορές, σε δόσεις μάλλον 500 φορές δυνατότερες ε, από ότι αυτές που δόθηκαν στους ανθρώπους. Πολλοί συμφωνούν πως αυτή η καταστροφή θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αν είχε χρησιμοποιηθεί η προηγμένη τεχνολογία των μικροδόσεων. Πάλι Πρόκειται για μια από τις εναλλακτικέ μεθόδους, όχι μόνο in vitro, όπως είπε σωστά η κυρία Ροτ Μπέρεντ. Υπάρχουν άλλες δυνατότητες και οι μικροδόσεις, μικροδοσολογία είναι μία από αυτές τις πιθανότητες. Προσπαθούμε λοιπόν να πιέσουμε τον κλάδο να χρησιμοποιεί όχι μόνο πειράματα υπάρχουν σήμερα, αλλά να δουν για παράδειγμα τι γίνεται και σε άλλους τομείς, όπως την μικροδοσολογία. Κυρία Μέρκο, παρακαλώ ολοκληρώσετε. Ναι, ναι, το ξέρω, θα, θα κλείσω. Πρόεδρος, μπορώ να σας ζητήσω να ολοκληρώσετε παρακαλώ, γιατί είναι πολύ ε, μακρύς, μακρά η ομιλία σας. Ναι. Μία τελευταία φράση. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ε, προηγμένες ε, εξελιγμένες ε, τεχνικές που μπορούν να επιτρέψουν ακριβή εξέταση των πιθανών πτώσεων στους ανθρώπους και θα ήθελα να τονίσω ότι δεν προτείνουμε το phase out στο, στα πρωτεύοντα εκτός από ανθρώπους. Δεν προτείνουμε το τέλος των ερευνών στην Ευρώπη, απλώς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εντός των οποίων η επιστήμη να ανθίσει, χωρίς νομοθετικά κίνητρα, κάτι τέτοιο δεν θα είναι δυνατόν. Αυτό είναι το κύριο μας μήνυμα. Το κύριο μας μήνυμα και στην επίσκεψη στο ΕΚΒΑΜ. Είπαν πως ήδη έχουν αναπτύξει και επικυρώσει εναλλακτικέ δοκιμές που δεν μπορούσαν όμως να χρησιμοποιηθούν διότι δεν επιτρέπονται από την νομοθεσία. Εμείς είμαστε οι νομοθέτες. Μια τελευταία παρατήρηση. Δεν υπάρχει... Δεν γίνονται αυτή τη στιγμή πειράματα για με τα μεγάλα πυθικοειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και καιρό δεν μπορώ λοιπόν να φανταστώ πώς και τι θα συμβεί σε περίπτωση μιας πανδημίας. Υπάρχει η διαδικασία 60 ημερών μέσω της επιτροπολογίας. Αν έχουμε μια πανδημία και έχουμε τα φάρμακα, πιθανότητα θα τα δώσουμε αμέσως σε εκατομμύρια ασθενείς. Και και δεν θα φτιάξουμε εργαστήρια για μεγάλα πυθικοειδή για να δοκιμάσουμε πρώτα. Η εντύπωσή μου είναι πως όλα αυτά είναι μια δικαιολογία. Γιατί ο δεύτερος λόγος για τον οποίο χρειάζεται αυτή η ρήτρα στο άρθρο 15 είναι πως, πως όλα αυτά χρειάζονται για την προστασία των ε, ε, ειδών ζώων που κινδυνεύουν το πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα αδέξιο ως επιχείρημα. Γι' αυτό και θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη της Επιτροπής ε, να σκεφτούν ότι είναι για μια καλή ευκαιρία ώστε να σταματήσουν αυτές οι ντροπιαστικέ δοκιμές, τα πειράματα, που δεν είναι καν απαραίτητα. με αυτή την πρόταση και κάποιες μικρές τροπολογίες εμείς οθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πιέζουμε αυτούς που υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνοι για να υπάρξει εξέλιξη. Χωρίς κάτι τέτοιο θα μείνουμε στο status κουβό που δεν είναι ικανοποιητικό. Jackson. Κύριε Τζάξον, για να διορθώσουμε κάτι, γιατί νομίζω ότι πρέπει. Η κυρία Μάρκο μας δημιούργησε την εντύπωση ότι υπάρχουν, ε, ότι γίνονται αυτή τη στιγμή κάποια ε, παρεμβατικά πειράματα ε, στα πρωτεύοντα, τα οποία δεν οδηγούν σε κανένα αποτέλεσμα. δεν είναι αλήθεια κάτι τέτοιο. υπάρχει θεραπεία για το Πάρκινσον που ονομάζεται ερέφισμα του εγκεφάλου. Γίνεται έγχυση ενός προϊόντος στον εγκέφαλο. Και εδώ θα ήθελα να ελεγχθεί σε ένα πρωτεύον και μετά σε μένα. Είναι πολύ αποτελεσματικό φάρμακο συμπεριλαμβάνει συνεχή έγχυση στον εγκέφαλο μια συγκεκριμένη ουσία. Έχει γίνει μια επίδειξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, Το διοργάνωσε το Ερευνητικό Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασίλειου. Το, το εν λόγω άτομο ε, στην ουσία ε, κατέρευσε. Ε, και στη συνέχεια έγινε φυσιολογικός, χωρίς, κανένα, ε, ε, χωρίς, χωρίς να τρέμει πλέον κτλ. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και δεν θα πρέπει να αφήσουμε αυτά τα οποία είπε η κυρία Μάρκο χωρίς να τα απαντήσουμε. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την κυρία Φερέρα γιατί πραγματικά μου ανέβασε το ηθικό. Yeah, Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τότε άλλη μια ανακοίνωση έχω να κάνω όσον αφορά τις ε, προθεσμίες για την κατάθεση τροπολογίων αύριο στις 10 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Και η τροπολογία στα αγγλικά σας παρακαλώ. Θα ψηφίσουμε στις 17 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια θα πάει στην Επιτροπή Γεωργίας, η οποία θα ψηφίσει στις 31 Μαρτίου. Εντάξει, ωραία. Τελειώσαμε λοιπόν τη συζήτηση για το θέμα αυτό και πάμε στο θέμα 6, προφορική ερώτηση του Chris Davis για τις ασιατικές αγριόγατες και τίγρες. Έχετε το λόγο κύριε Μπόρς. Δέβη, συγγνώμη. Uh, well, thank you, Chair, but, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτηση, την ερώτηση την έχουμε. Ε, θέλω να, ακούσω την απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνέχεια θα ήθελα να μου επιτρέπετε να το Namens Ωραία. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Λάγκεντροφ να τοποθετηθεί εκ μέρου τη Επιτροπή Περιβάλλοντο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία εμπεριέχονται στην ερώτηση. Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Υπάρχει μία ερώτηση που έχει να κάνει με το παράνομο εμπόριο των ειδών αυτών και το βαθμό στον οποίο η υφιστάμενη νομοθεσία εφαρμόζεται, καθώς και ορισμένες άλλες πτυχές. Ξεκινώ ε, με ορισμένα γενικά σχόλια για να τοποθετήσω το θέμα στη σωστή του Το διεθνές εμπόριο ε, τίγρης και προϊόντων τίγρης απαγορεύεται με βάση τη, τη σύμβαση ε, του Παγκόσμιου Εμπορίου ε, των επαπειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας στο λεγόμενο πίνακα 1. Δεύτερον, όσον αφορά το κυνήγι της Τίγρης απαγορεύεται και με βάση την εθνική νομοθεσία. Εδώ μιλάμε για χώρες όπως η Κίνα Ινδία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεύτερο, δεύτερη γενική παρατήρηση. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι στη συνδιάσκεψη των συμβαλόμενων ημερών στη Χάγη τον Ιούλιο του 2007 ενεκρίθη ένα ψήφισμα το οποίο καλούσε τα ενδιαφερόμενα μέρη, ε, τα, τα συμβαλόμενα μέρη της ΆΙΤΟΣ, να ε, πρώτα απ' όλα να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του λαθεμπορίου και του παράνομου εμπορίου. Ε, δεύτερον, να βελτιωθεί η περιφερειακή συνεργασία. Και τρίτον, να μην επιτρέπεται η εκτροφή σε αιχμαλωσία ε, ε, ε, της ε, τίγρεων για εμπορικούς σκοπούς. Τώρα τι έκανε η Επιτροπή για να υποστηρίξει προσπάθειες αυτές. Πρώτα απ' όλα η υποστήριξε δραστήρια το, ψήφισμα της Χάγης τον Ιούλιο του 2007. Ενέκρινε επίσης τον Ιούνιο του 2007 η σύσταση προς τα κράτη-μέλη όπου καθορίζονται μία σειρά από για τη βελτίωση ε, της εφαρμογής ε, της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθεσίας Άρητες και ζητά από τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν τις διεθνείς οργανώσεις, για παράδειγμα την Διεθνή Τελωνιακή Ένωση και την Ιντερπόλ. Βρίσκεται σε διαρκή επαφή άλλωστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις οργανώσεις αυτές και μάλιστα ε, όσον αφορά την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, που εργάζεται για το θέμα αυτό, ε, πρέπει να πω ότι συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Διεθνούς Τελωνιακής Οργάνωσης. Όσον αφορά την Κίνα και το τι κάναμε. Πρώτα απ' όλα, συζητήσαμε το θέμα αυτό με την Κίνα και σε διμερή βάση, αλλά και στα πλαίσια του Σάιτες, και ζητήσαμε ε, από την Κίνα να υποβάλει έκθεση στη μόνιμη επιτροπή. Πρώτα απ' όλα τον Ιούλιο του 2008 και στη συνέχεια τον Ιούλιο του 2009 να υποβάλει έκθεση για τις δράσεις που λαμβάνονται ως απάντηση στο ψήφισμα το οποίο ενεκρίθη ε, στη Χάγη. Χρηματοδοτήσαμε το 2005 ένα εργαστήριο στην Κίνα, ε, το εργαστήριο αυτό κάλυπτε την περιοχή της Ασίας, για τη βελτίωση, τη ε, συζήτηση και τη βελτίωση της ε, ε, συμμόρφωσης με την νομοθεσία και εδώ όσον αφορά το παράνομο εμπόριο και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η τίγρη. Θα το πράξουμε λοιπόν αυτό και φέτος θα το συζητήσουμε μαζί τους και γιατί χρηματοδοτούμε ένα εργαστήριο του σάιτες ειδικά για την τίγρη. Επίσης, έχουμε αναπτύξει ε, συγκεκριμένη ενημέρωση για το παράνομο εμπόριο επαπειλούμενων ε, ειδών, στην προκειμένη περίπτωση της τίγρης. Και εδώ συμμετέχουν ε, και εκπρόσωποι της παραδοσιακής ιατρικής στην Κίνα. Τώρα το κατά πόσο αναγνωρίζουμε, αυτή είναι μια άλλη ερώτηση το γεγονός ότι τα εγκλήματα στον ε, ε, τομέα των άγριων ζώων αποτελούν μια σημαντική μορφή του οργανωμένου ε, εγκλήματος, βεβαίως, ε, και εδώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την οδηγία, την αντίστοιχη οδηγία που αναφέρει συγκεκριμένα ότι είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως ποινικό αδίκημα το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων. Άρα λοιπόν ε, προβλέπεται και στην αδικία η ποινική δίωξη. Ένα άλλο ζήτημα είναι κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει οικονομική υποστήριξη στους διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται, όπως για παράδειγμα Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, η Παγκόσμια Οργάνωση Τελωνίων. Αυτή τη στιγμή δίνουμε ένα εκατομμύριο ευρώ σε σχέδια οικοδόμησης ε, ικανότητας από το site ε, στις χώρες αυτές και ταυτόχρονα προετοιμάζουμε τη δεύτερη φάση αυτών των σχεδίων οικοδόμησης ε, ικανότητας, πάλι ε, μιλώντας για εύρος ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ταυτόχρονα έχουμε και ορισμένα σχέδια περιφερειακής συνεργασίας με τη συγκεκριμένη περιοχή της Ασίας και εδώ καλύπτονται θέματα που έχουν να κάνουν με το, παρόμοιο, με το, με το λαθρεμπόριο και με την εφαρμογή του νόμου. Τέλο, όσον αφορά ε, το ρόλο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, πρέπει να σα πω ότι δεν γνωρίζουμε εμεί να υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα ε, ε, προς προ τι που να έχουν δημιουργηθεί από τι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Κυρίως το θέμα είναι εφαρμογή της εγχώριας νομοθεσίας στις εν λόγω χώρες. Δική τους ευθύνη λοιπόν είναι Και όσον αφορά τη δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσα να αναφέρω τι προσπάθειε τη Επιτροπή για να προωθήσει την ανάληψη κοινωνική ευθύνη ε, των συστημάτων ε, οικοδιαχείρισης και της πρόθεσης της συμμόρφωσης με τα μέσα του ΩΣΑ, όπως για παράδειγμα σε επίπεδο πολυμερών επιχειρήσεων, εξαγωγικών ε, ε, πιστώσεων και περιβάλλον. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να σταματήσω εδώ και να ε, ακούσω και τις δικές σας απόψεις. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες πολλών ε, ε, βουλευτών, ε, όπως επίσης ότι θέλει να προστατεύσει τα απειλούμενα είδη τα τίγρη προκαλούν ε, έντονα συναισθήματα. Μπορεί να μιλήσει κανείς για την απώλεια της βιοπικιλότητας, ε, η εξαφάνιση των ε, τίγρεων πάντως είναι κάτι που απασχολεί πολλούς ανθρώπους. Τρία πράγματα. Η Επιτροπή αναφέρθηκε στο ότι η Κίνα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να πετύχει κάποιους στόχους στα πλαίσια του site και το θέμα έχει τυχθεί και στο site και διμερώς με την Κίνα. Ε, η ερώτηση είναι λοιπόν ποια είναι η ανταπόκριση της Κίνας, ε, τι ε, εντύπωση δίνει η Κίνα σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλει για να πετύχει τους στόχους αυτούς της μείωσης δηλαδή της εμπορίας προϊόντων τίγρεως εντός της χώρας. Δεύτερον, ακούσαμε τι κάνει η Επιτροπή τι άλλο θα μπορούσε να κάνει η Επιτροπή, τι περισσότερο θα μπορούσε να κάνει ως προς την χρηματοδότηση, ως προς τις μεθόδους που ήδη αναφέρθηκαν, ως προς την ε, επιβολή των κανόνων παγκοσμίω. όσο τα αποθέματα, την ε, εξασφάλιση των τίγρεων σε σχέση με το παράνομο εμπόριο και επίσης τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει το Κοινοβούλιο για να βοηθήσει την Επιτροπή στις προσπάθειές της, για παράδειγμα ε, ανεβάζοντας το πολιτικό προφίλ του θέματος αυτού που είναι σημαντικό για τους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Ε, τον λόγο έχει η ε, Βαρόνι Λάτφορτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο παρότι δεν είμαι μέλος ε, της ε, Επιτροπής αυτής. Όπως είπε ο Κριστ Davis, τα... η τίγρης είναι ένα σύμβολο. Μ' αρέσουν οι μικρές και οι μεγάλες γάτες και εδώ και χρόνια ασχολούμαι με το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Πιο πολύ επαφή είχα ε, με την ε, περιβαλλοντική οργάνωση που βρίσκεται στην εκλογική μου περιφέρεια. Συνεργάστηκαν ε, με την Οργάνωση Προστασίας Άγριων Ζώων της, Κίνας, της Ινδίας και τύπωσαν ένα, ένα φυλάδιο το οποίο αναφέρεται στο γδάσιμο της γάτας πρόκειται για μια αγγλική έκφραση ότι μπορεί κανείς να γδάρει μια γάτα με πολλούς τρόπους ε, δεν είναι πολύ ε, ωραία έκφραση αλλά είναι επίγον το θέμα ε, η δυνατή εξαφάνιση της τίγρης είναι πρόβλημα και Είχαμε και άλλες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, είχαμε μια γραπτή δήλωση το 2006. Εγώ και άλλοι προβουλευτέ, ε, η Κομισιόν, του Συμβούλιο έχουμε καταβάλει διάφορες προσπάθειες. Ε, θα ήθελα να ε, σχολιάσω τις ερωτήσεις του Chris Davis ως προς την ανταπόκριση της Κίνας. Ένα πράγμα που τονίζουν οι εμπειρογνώμονες είναι η διατήρηση της απαγόρευσης στο εμπόριο προϊόντων τίγρεως εντός της Κίνας και στο κλείσιμο των εκμεταλλεύσεων ε, εκτροφής ε, τίγρεων, διότι υπάρχουν επενδυτές στον τομέα αυτών, 45.000 ε, εκτρέφονται στην ε, Κίνα. Τα επιχειρήματά τους είναι άχρηστα. Ε, θέλουν νομιμοποίηση του ε, εμπορίου, ε, αλλά ουσιαστικά θέλουν να εξοραίσουν τις δραστηριότητες τους, ε, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ε, επιβλαβής όσον αφορά την ε, διατήρηση των, ειδών, των τίγρεων. Ε, η Κομισιόν έχει συζητήσει το θέμα με την Κίνα. Η Κίνα είπε ότι είναι εσωτερικό θέμα, αλλά η, Κίνα είχε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε το θάρρος να θίξει απέναντι στην Κίνα το θέμα του κλεισίματος των ε, ε, εκμεταλλεύσεων εκτροφής ε, τίγρεων, διότι νομίζω ότι υπάρχουν πολλά κατεψυγμένα πτώματα τίγρεων σε καταψύκτες που στόχο έχουν να διατεθούν στην αγορά. Το 2007 η Επιτροπή απάντησε σε ερώτησή μου, είπε ότι ε, παρήχε στην Κίνα και στην Ινδία ε, τεχνική βοήθεια, αλλά ότι ε, το αρνήθηκαν, αυτό, αρνήθηκαν τη βοήθεια αυτή οι χώρες. Η Ινδία νομίζω ότι έχει συστήσει μια αρχή καταπολέμησης του του τον, το στον τομέα αυτών. Ε, η Επιτροπή έχει υποστηρίξει τις δραστηριότητε ε, της υπηρεσίας αυτής. Η, τρίτον, η Κομισιόν ε, θα μπορούσε να εξετάσει την προοπτική μιας ημερίδας ε, τίγρεων, ε, να ξεκινήσει δηλαδή μια συζήτηση ε, σε συνεργασία με άλλες χώρες, την Ινδία, την Κίνα κτλ. Έχουμε πολλά προβλήματα στον κόσμο, την απασχόληση, την, ε, τη διατροφική ασφάλεια, ε, λήψεις κλπ. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι το θέμα της διατήρησης της ε, βιοπικιλότητας είναι σημαντικό. Επίσης, μήπως θα μπορούσαμε να στείλουμε έναν πρέσβη, ειδικά για τις τίγρες στις χώρες αυτές. Είναι μια ιδέα που θα ενδιαφερόταν να προωθήσει η Κομισιόν. Ε, θα μπορούσε να είναι ένα δημοφιλές πρόσωπο, θα μπορούσε να είναι ε, κάποιος ηθοποιός του Bollywood ε, ή κάτι τέτοιο. Χρειάζεται φαντασία, χρειάζεται να πετύχουμε τη λαϊκή υποστήριξη στις χώρες αυτές για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες αυτές. Ε, δεν αρκεί η Δύση μόνο να υποστηρίζει την διατήρηση της ε, βιοπικιλότητας. Ε, θα ήθελα δηλαδή να προσθέσω στα ερωτήματα του Κρίς Ντέιβις. Τι ακόμα μπορεί να κάνει η Κομισιόν. Θεωρεί ότι κάνει αρκετά. Ευχαριστώ πολύ την Βαρόνι Λάτφορ. τον Τζον Μπόουις έχει το λόγο. Νομίζω ότι ε, μόλις έμαθα ποιος θα είναι ο ρόλος μου όταν εγκαταλείψω το κοινοβούλιο. Θα γίνω πρέσβης Τίγρεων. Θα ήθελα όμως ε, να θέσω μια σύντομη ερώτηση. Είναι σοβαρό θέμα. Το εμπόριο προϊόντων τίγρεων, τίγρεως με απασχολεί ιδιαίτερα. Ε, τέτοια προϊόντα χρησιμοποιούνται συχνά σε κινέζικα φάρμακα και σε άλλα προϊόντα. Πολλά από αυτά μπορεί να περνάνε σύνορα, να περνάνε τα Ιμαλάια, ε, για να παρακάμψει κανείς την αστυνομία, τα τελωνία κτλ. Πολλά από αυτά τα προϊόντα όμως πολλούνται και μέσω διαδικτύου και ε, ρωτώ την Κομισιόν τι κάνει για να έρθει σε επαφή με την Google και ε, άλλους φορείς για να ε, ε, πιάσει όσους έχουν ιστοσελίδες που διαφημίζουν τέτοια προϊόντα. Πώς μπορεί να ασκήσει η πίεση στην Google και στις άλλες τέτοιες επιχειρήσεις για να σταματήσουν την προβολή τέτοιων προϊόντων στις συστοθέσεις τους. Μπορούν να το κάνουν, γιατί το έχουν κάνει και σε άλλα θέματα. Ίσως έτσι θα μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε το εμπόριο μέσω διαδικτύου που κατά τα άλλα παρακάμπτει τις αρχές. Ευχαριστώ. Τζον Bowies ή Άβριλ Doyle. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα ε, προσεκτικά την απάντηση της Κομισιόν ε, και την ερώτηση του Chris Ντέιβις. Ενώ περιμένουμε την ομοθεσία που θα ακολουθήσει τις διαβουλεύσεις της Κομισιόν ε, για τα είδη αυτά, απελπίζομαι. Δεν πιστεύω ότι δίδεται προτεραιότητα στο θέμα αυτό, ούτε ότι υπάρχει πραγματική ανησυχία για θέματα βιοπικιλότητας. Μου φαίνεται ότι το όλο θέμα της βιοπικιλότητας και της έρευνας έχει πάρει τον κατήφορο Θα ήθελα η Κομισιόν να μου θυμίσει πώς ορίζει τα ξένα είδη. Διότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές ερμηνείας και με απασχολεί αυτό ιδιαίτερα ε, υπό το φως της αλλαγής του κλίματος. Είναι θέμα που θα συναντήσουμε. Θα συναντήσουμε θέματα προβλημάτων οικοσυστημάτων, ε, θέματα ε, ξένων ειδών, μη ηθαγενών ειδών. Ίσως η επαναπικοποίηση, η μεταφορά ειδών από τον νότο στο βορρά, ε, στις θάλασσες βλέπουμε αλλαγές ε, στα, στους τρόπους ε, αναπαραγωγής. Βλέπουμε ότι πολλά ψάρια μεταφέρονται στο βορρά λόγω της ε, θέρμανσης των θαλασσών. Βλέπουμε λοιπόν αλλαγές στα οικοσυστήματα πού ξεκινά και πού ε, κλείνει ε, το θέμα των ε, των ειδών. Η απεικιοποίηση, η αλλαγή του οικοσυστήματος, τα ξένα, είδα, τα ξένα είδη. Κυρία Ντόιλ, μήπως μιλάτε για το επόμενο θέμα. Νόμιζα ότι, μιλάμε, ότι συζητάμε και τα δύο μαζί, λέει η κυρία Ντόιλ μόνο για τις τίγρες μιλάμε. Συγγνώμη, ο, η, τίγρης, ε, η κέλτικη τίγρης ε, έχει πεθάνει. Δεν ε, ξέρω τι σχέση έχει με την παρούσα συζήτηση, αλλά εντάξει, μπορούμε να το εισάγουμε. Καλά, είπα αυτά που ήθελα. Ε, δεν ε, θα τα επαναλάβω κύριε Πρόεδρε αυτά που είπα, ε, απλά για να κλείσω το θέμα και ζητώ συγγνώμη. ο Γκρις ε, Τι θέση έχει στην Ευρώπη. Έχω βαρεθεί να ρωτάω την Επιτροπή. Ε, έχω κουραστεί να ρωτάω την Επιτροπή τι κάνει για τον Γκρι Σκίουρο που ε, απειλείται. Εάν συγκρίνουμε αυτά που κάνουμε για... Εάν συγκρίνουμε αυτά που κάναμε για τα εισβάλλοντα ήδη σε σχέση με αυτά που δεν κάναμε για τον Κρι Κύουρο, ε, κύριε Πρόεδρε, άχρηστα τα λόγια μας και ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μείνω στο θέμα της τίγρης και της ε, βιοποικιλότητας. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την τόσο πλήρη απάντηση που έδωσε στο ερώτημα του συναδέλφου Κρίς. Αλλά είναι αλήθεια ότι προσωπικά να σας πω ότι ήμουν εισηγήτρια για το σχέδιο δράση για τη βιοποικιλότητα και είναι αλήθεια ότι κάθε φορά που μιλάμε για ένα συγκεκριμένο είδος ε, και πολύ συχνά μιλάμε για επαπειλούμενα είδη και κοιτάξτε, ένα ε, είδος το οποίο αφανίζεται, αφανίζεται για πάντα. Πρέπει να καταβάλουμε λοιπόν κάθε προσπάθεια για να διατηρήσουμε τα είδη και κυρίως ε, ε, είδη όπως η τίγρης, τα οποία αποτελούν και την κοινή μας κληρονομιά, αν θέλετε. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις που θα ήθελα να θέσω όσον αφορά το τι κάνουμε εδώ στην Ευρώπη. Και αυτό συνδέθηκε με την ερώτηση του κυρίου Μπόβης. Μα είπατε ότι ε, αναγνωρίζεται ως μία μορφή οργανωμένου εγκλήματος και ότι ε, πρόκειται για πραγματικό αδίκημα. Μιλώ για αυτό το είδος του εμπορίου. Ρωτώ, εσείς ε, έχετε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά το εμπόριο αυτό στην Ευρώπη και έχετε, έχετε σε επαφή με τις διεθνείς με τη Διεθνή Οργάνωση Τελωνίων ε, όσον αφορά την απόκτηση στατιστικών στοιχείων. Και βεβαίως τώρα που έχουμε αυτές τις νέες μεθόδους αγοράς από το διαδίκτυο. Εδώ τι γίνεται, ε, όσον αφορά αυτή τη μορφή εμπορίου, έχουν στοιχεία τα τελωνία, μπορείτε να παρακολουθήσετε και αυτή τη μορφή εμπορίου. Ε, τώρα μας μιλήσατε για ένα εκατομμύριο ευρώ. Ε, και αναφερθήκατε σε αυτού του διεθνεί οργανισμού. Ηνωμένα Έθνη, Διεθνή Οργάνωση Τελωνίων. Κοιτάξτε, πριν από λίγα χρόνια ε, ήταν πιο σημαντικό το εμπόριο αυτό όσον αφορά κύκλο εργασιών σε σχέση με, τον, με το εμπόριο ναρκωτικών. Δεν ξέρω. Ε, καταλαβαίνω ότι γενικά υπάρχει οικονομική δυσκολία, αλλά αρκούν αυτά τα χρήματα. Το εμπόριο αυτό συνεχίζεται, μην το ξεχνάμε. Και έτσι κι σα ρωτώ, τι εκπροσωπεί το εμπόριο αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Υπήρου. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Αρχικά με ορισμένου συναδέλφου ε, μπήκαμε στον πειρασμό να φτιάξουμε ένα ψήφισμα για αυτό το θέμα, αλλά δυστυχώ δεν είχαμε χρόνο και χρειάστηκε να περιοριστούμε σε κάποιες ε, παρατηρήσεις. Θεωρώ πως είναι καλό ότι είμαστε πολύ δραστήριοι σε αυτό το θέμα. Πάντως στην Κίνα υπάρχουν ένα σωρό ε, <clears throat> εκμεταλλεύσεις αλλά και μαγαζιά που πουλούν τα ίδια αυτά χωρίς κανένα πρόβλημα. Κάναμε και μια ανακρόαση ε, για το θέμα αυτό. Είδαμε πως υπάρχουν πολλές ε, εκμεταλλεύσεις και πολλά καταστήματα γίνεται διάλογος ομαλά, αλλά στην πραγματικότητα δεν ε, σταματούν τίποτα. Ούτε πραγματοποιούν τις υποσχέσεις τους. Και έπειτα, τι κάνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείε για να μην υποβαθμίζουν το περιβάλλον. Όμως, το γεγονός είναι ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν είναι αυτές οι οποίες ε, βλάπτουν το σηκωτόπους των τίγρων, αλλά πολλά πράγματα συμβαίνουν παράνομα Πολλά γίνονται, καταστρέφονται τα οικότοποι των τίγρων. Οι τίγρες χρειάζονται μεγάλους ε, χώρους και δεν έχουμε τρόπο να εμποδίσουμε τα προϊόντα αυτά από τον άρθρο στην Ευρώπη. Γι' αυτό και θεωρώ πως ήταν και πολύ σημαντικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε ένα καλό μηχανισμό, μια καλή νομοθεσία και δουλεύουμε από αυτού. Και κάτι ακόμα, και εδώ κάνω έκκληση στην Κομισιόν, θα πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία για τις ε, συμφωνίες. Έχουμε υπογράψει μόνο μία. Έχω, το να υπογραφούν τέτοιου είδους συμφωνίες με την Κίνα ή την Ινδία βοηθά στο να λυθεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ja, dank u wel. Dan is nu het woord. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριο Ιούλιο Λάγκεντορφ. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα όσο μπορώ καλύτερα. Δεν είμαι βέβαιος πως μπορώ να τα ε, απαντήσω όλα, αλλά Νομίζω πως ε, το θέμα για τα εισβάλλοντα είδη θα είναι, για το είναι το επόμενο, γι' αυτό εκεί δεν θα απαντήσω τώρα. Η απάντηση που είχαμε λοιπόν από την Κίνα μέχρι στιγμή ήταν η εξή. Είχαμε μια πρώτη απάντηση σε σχέση με το ψήφισμα που εγκρίθηκε στην ΚΑΠ 14 στην Χάγη τον περασμένο Ιούλιο δεν θεωρήσαμε πως ήταν απόλυτα ικανοποιητική και γι' αυτό εμείς αλλά και άλλα μόνιμα μέλη αυτής της Επιτροπής ζητήσαμε από την Κίνα να μας αναφέρει και πάλι τι κάνει για το θέμα του ψηφίσματος στην επόμενη μόνιμη επιτροπή τον Ιούλιο του 2009. Ε, ε, πίεση λοιπόν ασκούμε στην Κίνα για να μας δώσει περισσότερες και πληρέστερες πληροφορίες για το τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει. Επίσης, ε, συζητάμε το θέμα αυτό με την Κίνα και στις διμερείς μας επαφές και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά την χρηματοδότηση, έχουμε κάνει ένα workshop που ιδιαίτερα, ειδικά αφιερωμένο στις Τίγρης. Ε, το πρώτο ήμιση του έτους, σε συνεργασία με την γραμματεία του Ε, προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε την οικοδόμηση ε, ε, δυνατοτήτων σε σχέση με το site τους. Προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε στη δεύτερη φάση για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς το θέμα των τίγριων. Τώρα υπάρχει και το θέμα του αν υπάρχουν άλλε πηγέ χρηματοδότηση. Εμεί στι ευρωπαϊκέ χώρε έχουμε καταστήσει σαφέ σε χώρε όπω η Ινδία πω αν το επιθυμούν μπορούν να εξετάσουν δυνατότητε χρηματοδότηση αλλά και ότι και ίδιοι πρέπει να κάνουν τέτοια αιτήματα για τα προγράμματα χρηματοδότηση. Αρκετές φορές έχουμε πει πως τέτοιου είδους χρηματοδότηση είναι δυνατή, αλλά πρέπει και εκείνοι να μας πούν από την άλλη πλευρά πως έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν επίσης. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχουμε διμερείς επαφές με την Ινδία και άλλες χώρες. Ε, προσπαθούμε να αυξήσουμε την ε, συνείδησή τους και την γνώση για το θέμα και να τους ε, καταστήσουμε επίσης γνωστό πως εάν το επιθυμούν μπορούν να έχουν και χρηματοδότηση σχέση, ανάλογα με τα προγράμματα συνεργασίας που έχουμε με την κάθε χώρα. διεθνές εμπόριο στα προϊόντα της τίγρης παραμένει απαγορευμένο. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Αυτό ισχύει εδώ και 34 χρόνια από τότε που υπογράφηκε η σύμβαση της Ουάσιγκτον. Το θέμα είναι βέβαια πως υπάρχουν, γίνεται μάλλον λαθρεμπόριο. Και έτσι έρχομαι σε ένα από τα ερωτήματα που ετέθησαν την κλίμακα δηλαδή του λαθρεμπορίου. Στον ΩΣΑ ζητήθηκε να γίνει μια μελέτη για τον εντοπισμό του αριθμού των των διαφόρων ειδών λαθρεμπορίου. Ένα είδος λαθρεμπορίου είναι και το εμπόριο αγρίων ζώων. Γι' αυτό και ζητήσαμε να γίνει έρευνα καταρχήν για να δούμε πόσο παράνομο, πόσο λαθρεμπόριο γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο και στη δεύτερη φάση θα εξεταστεί η δυνατότητα λήψης μέτρων, τα πιθανά μέτρα που μπορούν να ληφθούν στους διάφορους τομείς για να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο. Αυτή είναι μια από τις απαντήσεις λοιπόν που μας δόθηκαν. Τώρα για την παράνομη ξυλία στο βαθμό που σχετίζεται αυτό με το θέμα των τίγρεων. Έχουμε δουλέψει γι' αυτό. Εμείς ε, ε, συμμετέχουμε σε σχετικά προγράμματα. Ξέρετε επίσης και για τα, η πρότασή μας για την προσοχή που πρέπει να δοθεί. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε και σε σχέση με την Κίνα, όπου έχουμε αρχίσει διάλογο και για την παράνομη ε, δάσο, μάλλον υλοτόμηση των δασών. Θα γίνει τώρα και ένα διεθνές ε, σεμινάριο στον Καναδά αργότερα αυτό το μήνα, στο τέλος Φεβρουαρίου δηλαδή, που θα εξετάσει την πρόκληση του διεθνούς εμπορίου καθώς και με την ομάδα επιβολής θα περάσουμε μισή μέρα ακριβώς εξετάζοντας τις προσκλήσεις που ε, παρουσιάζονται λόγω του εμπορίου μέσω ίντερνετ. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι είναι πολύ θετικό το ότι εσείς μελετάτε με επίγοντα τρόπο το θέμα και ελπίζω να μπορέσουμε να σας δώσουμε περισσότερες απαντήσεις στον Ιούλιο που θα συναντήσουμε τα μέλη του Επιτροπής ΣΑΕΤΟΥΣ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λάγκεντορφ. Ολοκληρώνεται η εξέταση αυτού του θέματος εδώ και περνάμε στο ε, θέμα υπάρχουν 7. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Anne Teller, you have the floor. Κυρία Αν Τέλερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πότε κατάλαβα αυτό το θέμα ήταν μια προφορική ερώτηση που θα έπρεπε να απαντηθεί στην Ολομέλεια. Άδικο έχω. Όχι. Οπότε θα αφήσω την απάντηση της Κομισιόν για την Ολομέλεια. Αλλά ίσως προς χάρη διευκρίνησης για την κυρία Ντόιλα να πω ότι το θέμα των εισβαλών των ειδών έχει αναντοπιστεί από την Κομισιόν και έχει αναγνωριστεί ως ένα αυξανόμενο πρόβλημα στην Ευρώπη γιατί υπήρχε ένα κενό στην πολιτική μας για τη βιοπικιλότητα και γι' αυτό και υιοθετήσαμε μια ανακοίνωση στο τέλος του περασμένου έτους που αφορούσε τη νέα στρατηγική για τα εισβάλλοντα είδη. Εκεί αναφέρονται διάφορες επιλογές σε σχέση με τη στρατηγική της Ένωσης και τώρα έχουμε έρθει σε επαφή με διάφορα ε, θεσμικά όργανα, τα κρατημέλη, τους ενδιαφερόμενους φορείς και θα προχωρήσουμε με πρόταση για νέα στρατηγική για τα εισβάλλοντα είδη για το 2010. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Dank u σας ευχαριστώ. Η κυρία Τζάξον. Μια σύντομη ερώτηση προς την Επιτροπή. Δεν έχω καταλάβει καλά και με βάση αυτά τα οποία είπε ε, η Επιτροπή αλλά και με βάση την ερώτηση. Τι καλύπτουν τα εισβάλλοντα είδη, τα φυτά ή και τον αγαπημένο μας ε, κόκκινο σκίουρο. Βεβαίως εδώ δεν πρόκειται για εισβάλλον είδος, αλλά ρωτώ, υπάρχει ελπίδα να υπάρξει και κάποια οικονομική βοήθεια για την εξάλληψη ιδιαίτερα ε, ορισμένων ε, ε, ε που δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα στην νοτιοδυτική Αγγλία. Και στο Στρασβούργο παρατήρησα βέβαια. α, να, και, να, και άλλο ένα κακό με το Στρασβούργο. Και άλλη μια πληροφορία μάλλον που έχει να κάνει με το Στρασβούργο. Ποιος <coughs> ρωτώ ε, την ε, κυρία Τζάξον, μήπως εσείς το φέρετε στο Στρασβούργο ως μέρος της συνωμοσία κατά του Στρασβούργου. Όχι εντάξει, τώρα. Να πω το εξή. Αν περιμένουμε αυτό το 2010, τότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να έχει εξαφανιστεί τελείως ο σκύουρος αυτός. Ε, 120.000 είναι οι κόκκινοι και 3 εκατομμύρια οι γκρι Κάθε μέρα μειώνεται ο αριθμό των κόκκινων ε, ε, σκύουρων και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επιβεβαιώνει η Επιτροπή τι ευθύνε τη με βάση τη Σύμβαση για τη βιοποικιλότητα που αναφέρει ότι τα συμβαλόμενα μέρη θα παρεμποδίσουν την εισαγωγή θα ελέγχουν ή θα ε, μειώνουν ε, τα εισβάλλοντα είδη τα οποία απειλούν τα οικοσυστήματα, ζώα, φυτά κτλ. Πρέπει λοιπόν να ακούσουμε για τη δράση που έχει ήδη αναλυφθεί για την προστασία των ειδών. Και όχι απλά και μόνο να μιλάμε για το ότι θα φέρουμε νέες προτάσεις κτλ. σε ένα χρόνο. Εντάξει, μιλήσαμε για τους ε, ε και είναι σημαντικό το θέμα για την Ιταλία, για τη Γαλλία. Γιατί η τάση είναι από το Πιεμόντε να περνάει στη Γαλλία, η Βελβετία κτλ. Δηλαδή δεν περιορίζει το φαινόμενο ε, στη Βρετανία και στην Ιρλανδία. Υπάρχουν και πολλά άλλα είδη. Επίσης, ο σκόρος, που, ένα είδος σκόρου που καταστρέφει τις ε, βελανιδιές και που αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Ε, που προκαλεί άσθημα και αναφυλακτικό σοκ κτλ. Ε, αυτά τα πράγματα λοιπόν πρέπει να τα δούμε σοβαρότητα και να μας ανησυχήσουν και να κάνουμε κάτι. Και η Ευρώπη μπορεί συλλογικά να κάνει περισσότερα, διότι αυτά τα φαινόμενα είναι διασυνοριακά. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω λίγο περισσότερες πληροφορίες από την Επιτροπή για το τι γίνεται ήδη με βάση τη συγκεκριμένη σύμβαση. Καθώς επίσης να μας πει και δύο λόγια της προθέσης ε, της μέσα στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Κύριος Ντέβις, θα ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε ότι το θέμα αυτό το 7 ε, αφορά συγκεκριμένα το Συμβούλιο. Δεν είναι θέμα της Επιτροπής, είναι θέμα των κυβερνήσεων. Τα 27 κράτη-μέλη ε, στα οποία, ε, ε, ε, υπάρχουν τόσοι πολίτες και οι κυβερνήσεις έχουν συγκεκριμένες ευθύνες στο θέμα της βιοποικιλότητας και θα κάνουν τα επόμενα δύο χρόνια. Δηλαδή, θα ήθελα να ακούσω συγκεκριμένα στοιχεία. Πόσε φορές έχει συζητήσει το θέμα το Συμβούλιο, σε επίπεδο Συμβουλίου Περιβάλλοντος, γεωργία. Εδώ είναι αρμόδια πολλά Συμβούλια Υπουργών. Γιατί έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για μεγάλα λόγια και μεγάλες προσδοκίε που συμφωνούν στα λόγια τα κρατη και το αναβάλουν ε, για, μερικές, για μερικά χρόνια αργότερα. Είναι όπως όταν κανείς συμφωνεί να μιλήσει σε ένα, ε, σε ένα συνέδριο που νομίζω θα γίνει πολύ αργότερα. Λέει ναι βεβαίως και το ξεχνά. Ε, τελικά όμως κάποια στιγμή περνάει ο χρόνος και έρχεται η μεγάλη μέρα και αντιμετωπίζει την πραγματικότητα. Ε, αυτή την πραγματικότητα τώρα αντιμετωπίζει το Συμβούλιο. Μιλάμε εδώ για, την, για τον αφανισμό ειδών, ε, φυτών κτλ. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και το Συμβούλιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο. Ευχαριστούμε. Κύριε Ντόιλ, αν μου επιτρέπετε, να σα ευχαριστήσω για την υπομονή σα, κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω την Επιτροπή το εξή. Ποιο είναι ο ορισμό των εισβάλλοντων αυτών ειδών. και πού αρχίζει ε, η δημιουργία νέων απικιών λόγω της αλλαγής του κλίματος. Πώς κάνουμε διάκριση ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή, κοιτάξτε, Μπορεί να γελάμε με τον κόκκινο σκιούρο, αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα, παράδειγμα το οποίο το αντιλαμβάνεται όλοι εύκολα. Ε, αναφέρθηκαν και άλλα. Αναφέρθη, ε, η συνάδελφο αναφέρθηκε σε ορισμένα παράσιτα. Κοιτάξτε, η τεράστια καταστροφή στη βιοπικιλότητα και στα οικοσυστήματα αυτή τη στιγμή προέρχεται από χιλιάδες εισβάλλοντα είδη, τα οποία τυχαία ή εσκεμένα εισήλθαν στην Ευρώπη τον τελευταίο αιώνα. Και δεν ε, είναι αστεία όλα αυτά. Ανησυχώ γιατί πρέπει να περιμένουμε ένα-δύο χρόνια μέχρι να δούμε ένα σχέδιο πρόταση. Τουλάχιστον 18 μήνε λοιπόν με όλε τι καλέ προθέσει, ε, γνωμοδοτήσει, επιτροπέ, μέχρι να φτάσει στην Ολομέλεια. Άρα πιστεύω ότι εδώ μιλάμε για τουλάχιστον 4 χρόνια μέχρι να ληφθεί δράση στην Ευρώπη για το συγκεκριμένο θέμα. Και μετά, κοιτάξτε, δεν θα υπάρξει αναδρομική ισχύει. Ή το ξέρω διαφορετικά. Ερώτηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν επιτρέπεται αναδρομική εξέταση των περισσότερων ζητημάτων στα πλαίσια τη ε, νέου τη νομοθεσίας. Για παράδειγμα, θα υπάρξει δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το θέμα του κόκκινου σκιούρου ε, όταν θα έχουμε την νομοθεσία για τα εισβάλλοντα ήδη μετά από τρία χρόνια. Ή θα μιλάμε ε, γιατί θα γίνει από τα τρία χρόνια αυτά και μετά, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό θα γίνει, έτσι. Οι Ιταλοί πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα το θέμα του σκιούρου. Γιατί δεν θα έχουμε τελικά καρύδια για να βάλουμε στα Φεραίρο Ροσέ. Μα καταλαβαίνετε αυτό, όλα είναι ντροπή. Ε, ε, και, και τελικά ε, όλα αυτά έχουν καταστροφικές συνέπειες. Τεράστιες οικονομικές συνέπειες και ε, απώλεια από άψη βιοποικιλότητα που προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από αυτά τα εισβάλλοντα είδη σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και δεν το έχουμε αντιληφθεί, δεν έχουμε αντιληφθεί το θέμα, ε, πόσο σοβαρό είναι το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, προτείνω να τελειώσουμε τώρα με το θέμα αυτό τη ημέρης της διάταξης. Εδώ συζητάμε τι μεθόδου, διάφορε μεθόδου εδώ και 20 χρόνια και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα τι, ε, ε, να δούμε τι γίνεται. Για να δούμε. Ε, και πώς θα λύσουμε το θέμα για το σκιούρο. Προτείνω να ψηφίσουμε το οποίο θέλει να θέσει το θέμα αυτό στην Επιτροπή και ποιο θέλει στο Συμβούλιο. Ποιο θέλει την Επιτροπή, σηκώστε τα χέρια, εντάξει. Και ποιοι θέλουν να τεθεί το θέμα στο Συμβούλιο. Κατά. Κανείς. Ομόφωνα. Λοιπόν, ψηφίστε εποχή. Πάλι, πάλι, πάλι. Υπέρ, υπέρ. Τον ερωτήσε προς συμβούλιο. Ωραία. Ομόφωνα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να, ξε... ξεκαθαρίσω το εξή. Εμεί θεωρήσαμε ότι η συζήτηση αυτή κράτησε πάρα πολύ. Αυτό θέλω να πω και τίποτα άλλο. You are right. Um, Έχετε δίκιο. Επόμενο θέμα στη ημερήσια διάταξη. ε, σήμερα των ελαστικών πισώτρων αναφορικά με την οικονομία καυσίμου. Η συντάκτρια δεν είναι εδώ και θα ε, πάρει τη θέση της η κυρία Χάση. Täällä lyhyesti, koska todella aikaisemmat asiat ovat vieneet paljon aikaa. Tässä on kysymys autojen polttoaineen kulutuksen vähentämisestä, mutta... Χρειάστηκα πάρα πολύ χρόνο. Ε, υπάρχουν κάποιες πτυχές όμως που έχουν να κάνουν με τη μείωση της φθοράς, του θορύβου κλπ. Αυτή τη στιγμή η αγορά ελαστικών στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Οι καταναλωτές όμως δεν λαμβάνουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές στην απόδοση των διαφόρων ελαστικών. Έτσι λοιπόν η τιμή και ε, η φήμη της μάρκας ε, καθορίζει την επιλογή του καταναλωτή. Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή. Η 20 με 30% της ε, ενέργειας πρόθεση ενός οχήματος ε, σκοπό έχει ε, να ξεπεράσει την τριβή των ελαστικών και γι' αυτό υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην απόδοση ανάμεσα στα διάφορα είδη ελαστικών. Εάν η μέση τριβή όλου του στόλου των αυτοκινήτων ε, ε, βρισκόταν στο ε, επίπεδο των καλύτερων ελαστικών, θα είχαμε 5% μείωση στη χρήση των καυσίμων. Δηλαδή, ο καταναλωτής μέσα σε 5 μήνες θα είχε πάρει τα λεφτά του πίσω. Σκοπός μας λοιπόν είναι να ενημερώσουμε καλύτερα τον καταναλωτή, να ε, τον καταστήσουμε ικανό να ε, λαμβάνει ε, σωστές αποφάσεις με βάση σωστές πληροφορίες. Βέβαια, τα καλύτερα ελαστικά στον κόσμο δεν θα μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων εάν είναι κακή η συμπεριφορά των οδηγών. Ούτε μπορούν τα καλά ελαστικά να αντισταθμίσουν το γεγονός ότι κάποιες μηχανές αυτοκινήτων ε, καταναλώνουν πολλά καύσιμα. Η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών στον όσον αφορά τον θόρυβο και ε, την ε, αντιολυσθητική ικανότητα των ε, ελαστικών θα ήταν χρήσιμη. Οι τροπολογίες της Rebecca Harms σκοπό έχουν να ενισχύσουν την πρόταση της Κομισιόν και τους στόχους της, όπως για παράδειγμα στο θέμα του θορύβου. θα θα πρέπει να εισάγουμε ένα απλοποιημένο σύστημα, κάτι με ένα σήμα σαν φανάρι, διότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη σημασία των decibel. Οι τροπολογίες της Rebecca Harms επίσης ε, σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν την Κομισιόν να δημιουργήσει ιστοσελίδα όπου θα είναι διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα στοιχεία στους καταναλωτές. Αυτά κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Χάση. Ε, το λόγο έχει Μάρτιν Και εγώ θα προσπαθήσω κύριε Πρόεδρε να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Ε, η κυρία Χάση ε, επικεντρώθηκε στο θέμα της ε, απόδοσης των, στην εξοικονόμηση καυσίμων και στο θέμα του θορύβου των ελαστικών. Να μην ξεχνάμε όμως και την πτυχή της ασφάλειας. Θα πρέπει να μας απασχολεί, για παράδειγμα, η απόσταση που χρειάζεται για να φρενάρει κανείς όταν είναι βρεγμένα τα λάστιχα. Πάντως επικροτώ την πρόταση ε, άλλωστε τα λάστιχα τα αγοράζει κανείς από ανάγκη. Κανείς ε, δεν πάει για απλά καψόνια ε, για να αγοράσει ελαστικά. Ίσως το κάνει η κυρία Χάση, αλλά δεν νομίζω ότι κανείς άλλος το κάνει. Ε, σκοπός είναι λοιπόν η καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Κομισιόν σε κανένα δύο θέματα. Η Κομισιόν προτείνει υποχρεωτική επισήμανση των ελαστικών. Κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε ε, αν ε, ο κόσμος κοιτάει στο ράφι τα λάστιχα το ένα μετά το άλλο. ο κόσμος συνήθως κοιτάει τα λάστιχα σε καταλόγους, λαμβάνει πληροφορίες από τους πολίτες. Δεν είμαι βέβαιος λοιπόν αν είναι τόσο σημαντικό να έχουμε επισήμανση σε κάθε λάστιχο. Ε, εξίσου σημαντικό είναι οι σχετικές πληροφορίες να τυπώνονται στα ε, διαφημιστικά φυλάδια και σε άλλες μορφές. Ούτε με χαλά ιδέα της κυρίας Χάρμς ε, για τη δημιουργία ιστοσελίδας. Είμαι όμως ε, κατά της ε, πρότασης ε, να ε, κατηγοριοποιούνται με ενιαίο τρόπο τα χαρακτηριστικά. Είμαι υπέρ του να έχουν οι καταναλωτές όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες, δεν είμαι βέβαιος όμως εάν το κόστος του μέτρου αυτού του να τυπώνονται δηλαδή στο πλάι του λάστιχου, να εντυπώνονται ε, ανάγλυφα στο πλάι του λάστιχου όλες οι πληροφορίες, ε, δεν νομίζω ότι ε, αξίζει τον κόπο και ότι δικαιολογείται το επιπλέον κόστος. Αυτά κύριε Πρόεδρε είναι τα βασικά πράγματα που ήθελα να πω. Ε, προσλέπω στην όσο γίνεται πιο στενή συνεργασία με την κυρία Χάρμς για να έχουμε μια ισορροπημένη έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Μάρτιν Κάλανα, ο Ματίας Γκρότ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι σύντομος, λογικό βήμα αφού υιοθετήσαμε τον Δεκέμβριο την έκθεση Σακώνη. Τώρα έχουμε τα ε, συμπληρωματικά μέτρα, για παράδειγμα τη βελτίωση της ε, απόδοσης ε, των ελαστικών αυτοκινήτων. Πολύ σημαντικό είναι η ασφάλεια να προέχει, αυτό το ανέφερε ο προλαλής σας, ο κύριος Κάλαναν, και ε, παρέχεται η ασφάλεια αυτή με ε, τα μέτρα που προτείνονται. Αυτό ε, που είχαμε στην έκθεση Σακώνη ήταν τα νέα αυτοκίνητα. Τα, νέα αυτοκίνητα. τώρα όμως έχουμε μέτρα τα οποία θα ωφελήσουν και την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. θα Μπορεί δηλαδή να εξοικονομήσει κανείς σε καύσιμα και σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Κρίμα που δεν είναι εδώ η συγγήτρια, ήθελα να τη ρωτήσω κάτι, ίσως να μπορεί να μου απαντήσει όμως η ε, συνάδελφος Χάση. Στην ε, τροπολογία 18 γιατί υπάρχει διαγραφή. Ε, έχει διαγραφεί ολόκληρη σειρά και επίσης όσον αφορά την ιστοσελίδα έχω ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Κομισιόν σχετικά με το γραφειοκρατικό άχθο, ε, άχθος διότι ποιος θα πληρώσει για τη δημιουργία ιστοσελίδας. Θα παρακαλούσα την Κομισιόν λοιπόν να μου απαντήσει στο θέμα αυτό. Επίσης, ποια, ποιες είναι οι συνέπειες ε, της πρότασης αυτής ως προς ε, τη σκόνη που προκαλείται από την φθορά των ελαστικών. Ε, είχαμε μιλήσει για τα σωματίδια. Ε, θα παρακαλούσα την Κομισιόν λοιπόν να αναφερθεί στο θέμα αυτό. Επιπλέον θα πρέπει να σκεφτούμε εάν θα πρέπει να ε, είναι οδηγία ή κανονισμός ε, το συγκεκριμένο μέτρο. Θα ήθελα η Κομισιόν να μου εξηγήσει γιατί ε, προτείνει οδηγία και όχι κανονισμό. Ως προς την επισήμανση η κυρία... Η κυρία Χάρμς προτείνει τρία στοιχεία να αναφέρονται, εγώ πιστεύω θα πρέπει να αναφέρεται και η αντίσταση διότι ε, αυτό ε, είναι κάτι που παίζει ρόλο ως προς την απόδοση των καυσίμων. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να διατηρήσουμε απλά τα μέτρα, να μην κάνουμε πολύπλοκη την υπόθεση, ώστε ο κάθε καταναλωτής να μπορεί να μπει σε ένα κατάστημα ή από έναν κατάλογο να επιλέξει το καλύτερο λάστιχο. Γι' αυτό βρίσκω ότι αυτό που προτείνει η κυρία Χάμς, ιδιαίτερα καλό την επισήμανση για τα δεσιμπέλ. Ε, εάν αυξάνεται ο θόρυβος κατά 3 δεσιμπέλ, έχουμε διπλασιασμό του θορύβου. Αυτό το ξέρουν πολύ λίγοι, είναι λογαριθμική η αύξηση. Ε, γι' αυτό βρίσκω πολύ καλή την πρόταση της κυρίας Χάρμς να υπάρχει επισήμανση σαν φανάρι. Το τι μορφή θα έχει τελικά αυτή η επισήμανση θα πρέπει να το εξετάσουμε θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες και περιμένω αγωνίως να ακούσω τι θα μου απαντήσει η Επιτροπή. Και εγώ έχω μία παρατήρηση. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων Γενικά βάζουν φτηνά και κακή ποιότητα λάστιχα στα νέα αυτοκίνητα. Οι καταναλωτέ δεν το γνωρίζουν αυτό και δεν έχουν τι πληροφορίε που χρειάζονται για να διαμαρτυρηθούν κατά ε, αυτής της πρακτικής. Τελικά ο καταναλωτής ε, πληρώνει δηλαδή ε, περισσότερα καύσιμα και τα ε, λάστιχα φύρονται γρηγορότερα. Πιστεύω ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές. Ε, αυτό θα πρέπει να το καταστήσουμε θέση Η Κομισιόν έχει το λόγο. Η Κομισιόν θέλει να προσθέσει κάτι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, θα προσπαθήσω να επανέλθω σε ορισμένα σημεία. Καταρχήν ευχαριστώ την ε, κυρία Χάμζη για την εργασία της. Καθώ και για τη συζήτηση αυτήν την Επιτροπή για μια έκθεση που θα είναι χρήσιμη ιδιαίτερα όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργεια, αλλά και τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα και τις, εξ, για τον καταναλωτή. Ακούσαμε διάφορες ερωτήσεις ε, που ακόμα περισσότερες έχουν αναφερθεί στην έκθεση της κυρία Χάρμς αλλά ίσως κάποιες ε, ερωτήσεις τι οποίες να επανέλθω. Καταρχήν, για παράδειγμα, θόρυβος είναι ασφαλές πως πρόκειται για ενόχληση και για ενόχληση την οποία αξίζει τον κόπο κανείς να ασχοληθεί γιατί πιστεύουμε δύο άλλες παράμετροι που βρίσκονται στην ετικέτα και την οποία έχουμε παρουσιάσει είναι πιο σημαντικές για τον καταναλωτή δηλαδή η μείωση της κατανάλωσης και επίσης η ασφάλεια είναι πολύ ζωτική σημασία στα σημεία ενώ ο θόρυβος είναι ο θόρυβος τον οποίο ε, δημιουργεί το αυτοκίνητο για, εκτός του ίδιου του αυτοκίνητου. Δηλαδή είναι ο θόρυβος που προκαλούμε στους άλλους. Δηλαδή φοβόμαστε πως οι καταναλωτές δεν είναι τόσο ευαίσθητοι για το θόρυβο που προκαλούν για τους άλλους από τη στιγμή που ο θόρυβος δεν τους ενοχλεί στο εσωτερικό του αυτοκινήτου του. Φοβόμαστε επίσης ότι το να τονίσουμε περισσότερο το θόρυβο θα σημαίνει πως θα είναι εις βάρος της προσοχής που θα δώσει ο καταναλωτής στα δύο άλλα σημαντικά στοιχεία της ετικέτας και γι' αυτό πιστεύουμε όπως το προτείνουμε είναι μια καλή ισορροπία ανάμεσα στις δύο βασικές παραμέτρους ώστε να βελτιστοποιηθεί οι, οι δύο παράμετροι αυτοί χωρίς η μία να γίνεται εις βάρος της άλλης ενώ για το θόρυβο είναι μια πληροφορία την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επαγγελματίε, κυρίω για παράδειγμα όταν πρόκειται για δημόσιε προμήθειε, για κρατικέ δηλαδή αγορέ, όπου οι ίδιε οι αρχέ θα πρέπει να κάνουν ε, τι κατάλληλε επιλογέ, γιατί εκείνοι γνωρίζουν τον αντίκτυπο του θορύβου στο περιβάλλον. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι είχαμε πει για να γράψουμε κάποια στοιχεία στο πλάι των ε, ελαστικών. Πέρα από το κόστος που δεν είναι τεράστιο, το να μπουν δηλαδή πληροφορίες στο πλαϊνό μέρος του λάστιχου, πιστεύουμε ότι θα ήταν αντιπαραγωγικό γιατί ήδη πολλά πληροφορίε είναι γεγραμμένες πάνω στα λάστιχα και είναι πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή όταν θέλει να επαληθεύσει την ε, πίεση που είναι σημαντικό σημείο και για την κατανάλωση και για την ασφάλεια. Όσοι ήδη έχουν προσπαθήσει να δουν ποια είναι η πίεση στα λάστιχά τους, θα γνωρίζουν πως ήδη είναι δύσκολο να δείτε ποιο είναι το τύπος του ελαστικού που έχετε για να μπορέσετε να ε, διαπιστώσετε ποια είναι η κατάλληλη πίεση. Άμα βάλουμε και άλλα περισσότερα στοιχεία πάνω στο λάστιχο, θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο. Είναι μια πληροφορία λοιπόν που δεν είναι πραγματικά Υπάρχουν επίσης ερωτήσεις σε σχέση με το γεγονός ότι τα ταξινόμηση που έχουμε παρουσιάσει περιλαμβάνει και μια κοινή θέση. Μπορώ να καταλάβω την ε, απορία διαφόρων, το έχουμε ήδη εξηγήσει. Στόχος είναι βασικά να δημιουργηθεί ένα εφέ, κάπως τεχνητό εφέ, όπως ε, ναι όντως θα είναι τεχνητό, αλλά για να πιο προφανής η διαφορά απόδοσης στις ετικέτες για τον καταναλωτή. Πιστεύουμε δηλαδή ότι αν τα πράγματα είναι πιο θεαματικά, ας πούμε, έτσι, αν έχουμε δηλαδή και ένα κενό και μια κοινή θέση, ο καταναλωτής θα έχει να κάνει μια επιλογή ξεκάθαρη. Δηλαδή θα λέει είτε θα πάρω το λάστιχο στο καλύτερο επίπεδο, είτε θα πάρω το λάστιχο που έχει χαμηλότερες επιδόσεις. Και το γεγονός ότι υπάρχει μεγαλύτερη διάκριση, δηλαδή αν υπάρχει μεγαλύτερο κενό ανάμεσα στο πρώτο και στο καλύτερο και στο χειρότερο, Πιστεύω πως αυτό θα αναγκάσει τον καταναλωτή να επιλέξει τις καλύτερες κλάσεις, γιατί διαφορετικά μπορεί να υπάρξει αποδυνάμωση των ε, κλιμάκων αυτών. Κάπως πιο θεματική να είναι η ταξινόμηση δηλαδή για να πιέσουμε, να, να οθήσουμε μάλλον τον καταναλωτή να επιλέξει πιο ψηλά επίπεδο ποιότητας. Κάτι ακόμα που έχουμε τονίσει είναι το γεγονός ότι τα χειμερινά λάστιχα δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την πρόταση. Όντως είναι πολύ εύστοχη αυτή η παρατήρηση του εισηγητή και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι η ιδέα του να ορίσουμε τις λεπτομέρειες μέσω της επιτροπολογίας θα ήταν μια προσέγγιση έγκυρη. Ε, έπειτα, ένα σημαντικό στοιχείο επίσης που αναφέρθηκε στην έκθεση είναι τα αναγωμωμένα επίσωτρα. Δηλαδή είναι εκείνα τα κομμάτια ελαστικού που προστίθενται στα άλλα ελαστικά και που δεν καλύπτονται εδώ. Εμεί θεωρήσαμε πω ήταν καλύτερο να μείνουν εκτό του πεδίου εφαρμογή για την ώρα. Από τη μια πλευρά, γιατί δεν υπάρχει ακόμα μέθοδο μέτρηση που θα επέτρεπε να τα συμπεριλάβουμε και να τα ταξινομήσουμε και άρα να εποπτεύουμε και τη δήλωση του κατασκευαστή. Έπειτα θα πρέπει να γνωρίζουμε πω η απόδοση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το συνδυασμό του αρχικού λάστιχου με την ε, αναγόμωση που θα το γίνει. Υπάρχουν ένα σωρό δυνατότητες συνδυασμού. Σε κάθε συνδυασμό πρέπει να κάνουμε έλεγχο και εκεί το κόστος γίνεται απαγορευτικό. Για μια επιμηχανία που βασικά πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, κινδυνεύουμε να σταματήσουμε μια, έναν κλάδο που σε περιβαλλοντικό επίπεδο είναι ευεργετικός. Γιατί για κάθε αναγόμωση που γίνεται σημαίνει πως δεν χρειάζεται να ανακυκλωθεί αυτό το λάστιχο. Δηλαδή ο απολογισμός περιβαλλοντικός είναι θετικός όταν μιλάμε κυρίως και για τα βαριά οχήματα. Γι' αυτό για την ώρα προτιμήσαμε να μην το βάλουμε στην πρόταση. Πράγμα που δεν εμποδίζει βέβαια σε μια αναθεώρηση της οδηγίας να προβλέψουμε να εισάγουμε την αναγόμωση. Να μην τα αποκλείουμε δηλαδή από το πεδίο εφαρμογή αργότερα. Κάτι επίση που αναφέρθηκε στην Επιτροπή Ήτρε ήταν ότι Μπορεί να δοθεί εντύπωση πως η Κομισιόν κάπως τρελάθηκε, θέλει να βάζει ετικέτες παντού και κυρίως ε, πάνω σε κάθε ένα ε, λάστιχο. Θα πρέπει να γνωρίζετε πως ούτως ή άλλως υπάρχουν ετικέτες για όλα τα λάστιχα και που υποδεικνύουν τα κυρία χαρακτηριστικά του λάστιχου, για παράδειγμα τις διαστάσεις του και πράγμα που επιτρέπει σε όσους χειρίζονται αυτά τα λαστικά να ξέρουν για ποιο λάστιχο είναι και να μην χρειάζεται να διαβάσει και να αποκρυπτογραφήσει τα τα πλευρά, τις πλαϊνές πλευρές του ελαστικού. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι κάπως να μεγαλώσουμε αυτή την ετικέτα για να βάλουμε και αυτή την πληροφορία. Δηλαδή δεν πρόκειται να ξαφνικά να αρχίσουμε να βάζουμε ετικέτες σε κάθε ελάστιχο. Επίσης πιστεύουμε πως είναι ο μόνος τρόπος να εγγυηθούμε την ύπαρξη των πληροφοριών αυτών, τη διάθεση αυτών των πληροφοριών, για να ε, προσελκύσουμε την προσοχή των εμπόρων αλλά και των πελατών όταν προβαίνουν στην αγορά ελαστικών. Και όπως το είπε και ο κύριος βουλευτής, πρόκειται και για λάστιχα αντικατάστασης που είναι πάνω από τα τρία τέταρτα της αγοράς ελαστικών. Υπάρχει λοιπόν, έχει νόημα μια τέτοια πρόταση. Αυτά λοιπόν, αν έχετε και άλλες ερωτήσεις μπορώ να επανέλθω. Ευχαριστώ. Dan is het woord σας ευχαριστώ κύριε Χάση. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και την Επιτροπή για τις απόψεις σας. Τώρα, ε, προφανώς ε, δεν μπορώ να ε, μιλήσω για όλα τα θέματα για λογαριασμό της Ρεμπέκα Χάρμς. Θα τις μεταφέρω όμως αυτά τα οποία είπατε. Όσον αφορά το ζήτημα των ε, ε, πληροφοριών ε, επάνω στο, στο ελαστικό, καταλαβαίνω ότι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι μάλλον, το κόστος είναι ελάχιστο. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε, το, το κόστος θα, ήταν ε, ε, απαγορευτικό. Πραγματικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όσον αφορά την κατηγορία D, Εδώ να σας πω ότι συμφωνώ με την εισηγήτρια και εφόσον ε, έχουμε αυτή τη σήμανση ε, που έχει να κάνει με τα καταναλωτικά αγαθά και οι άνθρωποι καταλαβαίνουν συγκεκριμένα τι υποδηλώνει το α, το β, το a, το b, το c. Τι θα γίνει με το D, θα είναι κενό με το Δέλτα, με την κατηγορία Δέλτα. Κοίταξε για παράδειγμα, ε, ε, ε, στα, στα καταστήματα φαίνεται όσον αφορά τα ψυγεία ότι το α είναι το καλύτερο. Και όμως το καλ... δεν είναι το α, γιατί δε, ε, στα, στα καταστήματα δεν υπάρχει το α συν και το α2 συν. Όσον αφορά λοιπόν τη σήμανση πρέπει να είστε πιο συνεπείς. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, χρονοδιάγραμμα ε, για κατάσταση τροπολογιών 11 Φεβρουαρίου το μεσημέρι στις 12 η ώρα θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος 16 Μαρτίου και προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στην Επιτροπή Βιομηχανίας 24 Φεβρουαρίου και ψηφοφορία στην Επιτροπή Ήτρε 30 και 31 Μαρτίου και θα ζητηθεί στην Ολομέλεια του Μαΐου του 2009. Ε, τώρα ζητώ από την κυρία Χάση να αναλάβει την Προεδρία. No niin, hyvät ystävät Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ένα θέμα έχει μείνει. Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα. Συντάκτη Άννα Φερέρα που έχει και το λόγο. Oui, euh, Σας ευχαριστώ κυρία Χάση. Λυπάμαι που δεν έχουμε καθόλου χρόνο να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο έχω την εντύπωση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρόλο που η Επιτροπή μα ε, ε, γνωμοδοτεί απλά. Αυτή η ενωμένη κοινωνική ατζέντα είναι κάτι που την περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό και έρχεται καθυστερημένα. Και βεβαίω ε, περιέχει ορισμένα στοιχεία θετικά, αλλά ταυτόχρονα εκφράζουμε τη λύπη μα για το γεγονό ότι ε, παρουσιάζει ορισμένε ελλείψει που θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω την άποψη ότι τώρα περισσότερο από ποτέ έχει την υποχρέωση, ακριβώς αυτή τη στιγμή της οικονομικής κρίσης και της κοινωνικής κρίσης, να ε, δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια που αντιμετωπίζουν πάνω από 70 εκατομμύρια πολίτες και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες προσδοκούν μια Ευρώπη που να τους προστατεύει και να τους εξασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον ε, από κοινωνική άποψη αλλά και από άποψη περιβάλλοντος καθώς επί... μια καλύτερη ζωή και από άποψη υγείας. Ε, είμαι εισηγήτρια για την Επιτροπή μας για το θέμα αυτό ε, και μέσα στις ε, λίγες γραμμές που συνέταξα προσπαθώ να επικεντρώσω την προσοχή μας στα θέματα της υγείας και του περιβάλλοντος γιατί θεωρώ ότι είναι ο φτωχός συγγενής αν θέλετε τα δύο αυτά ζητήματα της πρόταση Επιτροπής. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσει τα σημεία αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι γνωρίζουμε ότι οι πιο ευαίσθητοι πολίτες είναι συχνά αυτοί που ε, εκτίθενται περισσότερο από τους υπόλοιπους σε ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον και δυστυχώς είναι οι ίδιοι που συχνά έχουν, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα υγείας. Επιμένουμε λοιπόν στα σημεία αυτά. Ε, ταυτόχρονα θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα θα πρέπει να συμπεριλάβουν, τα, τα, ε, να, να ε, ε, ε, δουν το θέμα ε, των σχεδίων για το περιβάλλον και την υγεία όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί της ουσίας, αυτό το έχουμε ξαναπεί εξάλλου επί της ουσίας θα πρέπει να υποβληθούν νέες προτάσεις που να αφορούν ακριβώς το θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επιπτώσεων μάλλον του περιβάλλοντος στην υγεία κάνοντας τη σύνδεση με τις διάφορες ασθένειες που, ε, στις οποίες εκτίθενται οι Ευρωπαίοι και εδώ αναφέρομαι συγκεκριμένα στην αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων καρκίνου. Κάτι άλλο το οποίο επίσης είναι σημαντικό είναι να δούμε με ποια μέσα μπορούμε να απαντήσουμε με τον καλύτερο τρόπο σε αυτά τα ερωτήματα τα περιβαλλοντικής φύσεως και ε, υγείας, να απαντήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης να δούμε τι γίνεται και σε επίπεδο δημοσίων υπηρεσιών. Βλέπουμε σήμερα ότι στην περίοδο κρίσης οι πολίτες στρέφονται προς ε, τη δημόσια εξουσία. Σήμερα έχουν καταλάβει οι πολίτες ότι οι απαντήσεις δεν θα έρθουν μόνο από τα κράτη-μέλη. Άρα προσδοκούν και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένες απαντήσεις όσον αφορά τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία αλλά και την ποιότητα της απασχόλησης πάντα σε σύνδεση με το περιβάλλον και με την υγεία. Και εδώ οι δημόσιες υπηρεσίες όπως και η κοινωνική οικονομία, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης της επασχόλησης, εδαφικής συνοχής, κοινωνικής συνοχής επίσης και νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στο σημείο αυτό. Και το έκανα και στην ε, ε, και στην γνωμοδότησή μου. Πρέπει να προωθήσουμε τόσο τι δημόσιες υπηρεσίε, υπηρεσίε υπηρεσίες κοινής αλλά και την, ε, κοινωνική οικονομία που παίζει σημαντικό ρόλο κυρίω στο θέμα τη υγεία. Ένα παράδειγμα θα αναφέρω για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Στα νοσοκομεία. Ε, στα νοσοκομεία θερα, ε, αντιμετώπισης των ε, περιπτώσεων καρκίνου για κάθε υπάλληλο του νοσοκομείου, για κάθε μέλος του προσωπικού έχουμε δύο θελοντές ε, αυτό γίνεται στη Γαλλία, αλλά φαντάζομαι ότι κάτι παρόμοιο γίνεται και σε άλλα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν όλοι να αναγνωρίσουμε τη σημασία όλων αυτών των θέσεων απασχόληση, που είτε αμείβονται δεν αμείβονται, είτε είναι θελοντικέ είτε όχι υπηρεσίε αυτέ, μέσα από τι οργανώσει, ε, τι οργανώσει αλληλοβοήθεια, διότι όλα αυτά ε, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο αναγνώριση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προθεσμία για τι τροπολογίε ε, προβλεπόταν για σήμερα σε 6 ώρα στην, αναβλήθηκε όμως για την Τετάρτη σεξ το απόγευμα και εγώ ίδια έχω προτείνει κάποιες διευκρινήσεις γιατί καταλαβαίνετε όταν κανείς πρέπει να γράψει 10 προτάσεις και μόνο για ένα θέμα ε, πρέπει να ασκήσει μεγάλη αυτό Και δεν ήμουν ιδιαίτερα διεξοδική κυρίως όσον αφορά τα ζητήματα υγείας. Πρέπει να αναφέρουμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ε, ποιοτικέ υπηρεσίες περίθαλψης κοντά στον τόπο στον οποίο διαμένει και η οδηγία ε, για, τις, ε, για τη διασυνοριακή περίθαλψη σίγουρα δεν λύνει το σύνολο των προβλημάτων αυτών. Αυτά όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει η έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Φεραίρα, πράγματι δεν έχουμε χρόνο. Οπότε, αν θέλετε το λόγο, συνάδελφοι, παρακαλώ να είστε πάρα πάρα πολύ σύντομοι. Προσπαθήσουμε να βρούμε λίγο χρόνο για να συζητήσουμε το θέμα ουσιαστικά. Αλλά αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και από το κατά πόσον θα έχουμε τη 16η Μαρτίου για την έγκριση αυτή τη γνωμοδότηση. Ο κύριο Μπούσελ Μάθιου θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Τέσσερι τροπολογίε που, πρόλαβα να τι υποβάλω πριν από 37 λεπτά. Τώρα όμω βλέπω ότι έχουμε αναβολή. Ελπίζω να καταλάβει η συγγητρία ότι η πρόθεσή μου είναι να σα βοηθήσω να ενισχύσετε την έκθεση. Δεν θέλω να την υπονομεύσω οι τρει τροπολογίε είτε προσθέτουν είτε αφαιρούν μία λέξη. Γιατί νομίζω ότι ορισμένε από τα σχόλιά σα, κατά την κρίση μου, είναι πολύ έτσι ξεκάθαρα χωρί αποχρώσει. Για παράδειγμα, στο Δέλτα, εκεί όπου αναφέρεται στην, ε, ε, στις σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές ε, ε, κρίσεις και το πώς επιδρούν όλα αυτά στο περιβάλλον και στο κλίμα. μπορεί να, προσθέτουν, να προσθέτουν αυτά στην κρίση, αλλά μπορεί και να μην προσθέτουν, γιατί λιγότερη βιομηχανική δραστηριότητα σημαίνει λιγότερη ρήπανση κτλ. Μια άλλη όψη του νομίσματος. Άρα να βάλουμε may add, ενδεχομένως να προσθέτουν. Έτσι, προτείνω ορισμένες αλλαγέ. Αλλά η τελευταία μου παρατήρηση έχει να κάνει με την παράγραφο 5. Εκεί όπου προτείνω, με όλο το σεβασμό, τη διαγραφή της. Όχι γιατί διαφωνώ, αλλά γιατί νομίζω ήταν καλύτερο αν υποβληθεί ω τροπολογία στην Επιτροπή σε απευθεία στην εισήγηση Σίλβα ε, ε είμαι εισηγητή ε, στην Επιτροπή αυτή και ασχολήθηκα με την αστυνομιακή υγεία ε, και εκεί είπαμε να μην έχουμε παρέμβαση στην έκθεση Boys για την περίθαλψη, εκεί όπου αναφέρεται οι κοινωνικές υπηρεσίες, ο ρόλος κοινωνικής οικονομίας, τη δημιουργία απασχόληση. Μα αυτό είναι ο κόσμο τη απασχόληση κοινωνικών υποθέσεων. Αν θέλετε λοιπόν κατευθείαν να πάει στην Επιτροπή Απασχόληση και είμαι σίγουρο ότι θα γίνει αποδεκτή. Σα παρακαλώ σκεφτείτε τι παρατηρήσει μου. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Συγγετρία. Σε γενικέ γραμμέ εκφράζει η Επιτροπή την ικανοποίησή τη για το σχέδιο έκθεση. Ίσως αν μου επιτρέπετε να επανέλθω σε δύο ή τρία σημεία τα οποία αναφέρονται στην έκθεση αυτή. Πρώτα απ' όλα αναφέρεται το ότι έχετε κάπως καθυστερημένη ανακοίνωση τη Επιτροπής αναφέρεται ε, τη σύνδεση με την οικονομική κρίση. Πράγματι να υπενθυμίσω ότι η ανακοίνωση αυτή ανακρίθηκε από την Επιτροπή τον Ιούλιο 2008, πέρυσι και τότε οι οικονομικέ συνθήκε δεν ήταν καθόλου ίδιες με αυτές ε, που υφίστανται σήμερα. Έπρεπε στο μεταξύ να απαντήσει στην οικονομική κρίση με το σχέδιο οικονομική ανάκαμψη που ενεκρίθηκε τον Νοέμβριο η Επιτροπή και που στη συνέχεια ενεκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εξάλλου, ως απάντηση στην οικονομική κρίση ε, θέλησε να συμβάλλει ουσιαστικά ε, στο προβληματισμό ε, και του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ε, όπου βεβαίως θα συζητηθούν ιδιαίτερα οι πτυχές που έχουν να κάνουν με την απασχόληση. Επίσης, να σας πω ότι σημειώνουμε μάλλον την ε, ε, ε, υποστήριξή σας στην ολιστική προσέγγιση. Βεβαίως, η απάντηση στις κοινωνικές προκλήσεις απαιτούν την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων πολιτικών και όχι μόνο τους. Της κοινωνικής εδώ, όπως σας παραπέμπω, στην πολιτική παιδείας, έρευνας, οικονομίας, περιβάλλον κτλ κοινωνία πληροφορία κτλ. Επίση, αναφέρεστε στην, καλύτερη ολοκλήρωση τη αηφόρων ανάπτυξη με τη Σαρδικής Λισαβόνα, βεβαίω, συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο πλαίσιο των ε, νέων στρατηγικών Λισαβόνα δηλαδή 2010 θα τα συμπεριλάβει όλα αυτά, ε, καθώ επίση και θα δούμε με ποιο τρόπο ε, μπορούμε να πετύχουμε τα μέλη στα αποτελέσματα. Αυτά ήθελα να σα πω σε γενικέ γραμμέ. Μια τελευταία παρατήρηση όσον αφορά αυτό το, το πρασίνισμα της ευρωπαϊκής οικονομίας, greening of the economy. Είναι και δική μας ανησυχία, και, αλλά θα πρέπει να δούμε και τις κοινωνικές επιπτώσεις και την πτυχή Αναπροσδιορισμό των δομών απασχόληση. Εργαζόμαστε προ την κατεύθυνση αυτή με στόχο να υποβάλουμε συγκεκριμένε προτάσει μέσα στου προσεχεί μήνε. Αυτά θέλω να πω και ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ την, Επιτροπ... την... τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. χρονοδιάγραμμα ως εξή. Προθεσμία saatiin, äh, saatiin keskiviikkoon kello 18 asti ja äh, päätös... Κοιτάξτε, όσον αφορά την προθεσία για τι τροπολογίε, Τετάρτη, 6 το απόγευμα, είπαμε, Και αν καταφέρουμε να έχουμε μια συνάντηση 16 Μαρτίου, τότε θα εγκρίνουμε την ε, γνωμοδότηση. Συναντήσει την περίπτωση στι 16-17 Φεβρουαρίου. Από ό,τι μου λέει όμως η γραμματεία, ε, ισχύει η 16 Μαρτίου. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Λίγη συνεδρία για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στην διεύθυνση.